Αγαπητοί συναδελφοί, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Και επαναρχόμεθα σε μια σειρά ψηφοφοριών. Πρώτα απ' όλα έχουμε πέντε γνωμοδοτήσεις για διάφορα προγράμματα, νομοθετικά προγράμματα. Ε, στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 21-27. Έτσι, νόμι είπα 5, στην ουσία είναι 4. Α, αλλά στην πραγματικότητα 3. Γιατί ο κανονισμός κοινών προβλέψεων έχει αναβληθεί. Πρώτη ψηφοφορία. Έκθεση Ούρμα το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. 30 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Με συγχωρείτε, αλλά δεν βλέπω πώς ψηφίσετε Υπέρ παρακαλώ ποιοι είναι. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 31 υπέρ κατά δεν είναι σαφές δεν είναι σαφές να ελέγξουμε την 31 άρχεται 31 σας παρακαλώ ψηφίστε ψηφίστε βάλτε τις κάρτες στο μηχάνημα ψηφίσατε όλοι από ό,τι φαίνεται όχι. Πέρας. Δεκτή. 13 υπέρ, 10 κατά. 32 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 3 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την τρία. άρχεται ψηφίσατε όλοι πέρας δεκτή 12 υπέρ 11 κατά Τέσσερα, πέντε και έξι. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές δεκτές 34 36 37 υπέρ Α, καταπίπτει, καταπίπτει, γιατί νεκρήθησαν οι 4-5-6, μάλιστα. 7, υπέρ. 7 λέω. Κατά. Ελέγχουμε την 7. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 13 υπέρ, 12 κατά. 8, 9, 10 και 11 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Άποχες. Να ελέγξουμε. Τις τροπολογίες 8 έως 11. Άρχεται. Πέρασε. 12-12. Απορρίπτονται. 39. Υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. 39. Ελέγχουμε. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ισοψηφία 12. Απορρίπτονται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Έλεγχος τις 14. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Απορρίπτεται. 11-13. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Την 15. Άρχεται. Πέρασε. Δεκτή 13-12. 16 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 17 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε. Την 17. Πέρας. Απορρίπτεται. 12-13. 18 υπέρ. Δεν αλλάζει τίποτα και με ισοψηφία 13 και πάλι απορρίπτεται. Έχουμε περάσει στην 18. 18 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 19 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά να δούμε ελέγχουμε την 22 ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται 21 υπέρ κατά με συγχωρείτε. Ε, να επανέλθω. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Την 24. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Μία ψήφος διαφορά. 13-14. Ήμασταν στην 24. 23 τώρα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Να ελέγξουμε την 23. Πέρας. 14, δεκατέσσερα. Αλλά απορρίπτεται λοιπόν. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχο, 25. Πέρας. Απορρίπτεται. 14-14. 26 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 26. Πέρας. 14-14. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 29 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Δεκτή, 25 υπέρ, 2 κατά και μία αποχή. Συγχαίρουμε τον ε, εισηγητή. Έκθεση John Howarth. Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Από κοινού 13, 14, 15, 16. Υπέρ Κατά. Αποχές δεκτές. Οι τροπολογίες. 3, 4, 5, 6 έχουν αποσυρθεί ή 7 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. σημαστική 1 υπέρ Κατά αποχές δεκτή. 2 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Η 12 έχει αποσυρθεί. Το σύνολο του κειμένου ονομαστική άρχεται. Δύο κάρτες δεν μπαίνουν στα μηχανήματα. Εντάξει, δεν με πειράζει εμένα. Πέρασε. Δεκτή, εγκρίνεται λέει το κείμενο 24-4. Ε, ε, Συγχαίρομαι τον κύριο Χάουαρθ. Τώρα θα περάσουμε στη θέση του Ταμείου Σύλλου και Μετανάστευσης, ε, έκθεση Καρίν Κλονέκ Μωρά. Επτά υπέρ. Κατά. Εποχές. Επαλήθευση ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 15 υπέρ, 13 κατά. 34 υπέρ, κατά. Εποχέ, απορρίπτεται. Τροπολογία 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 36, 50, 52, 56, 59 και 60 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη. Εγκρίνεται. 17 υπέρ, 11 κατά. Τώρα, τρεις τροπολογίες, 4, 5 και 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 37 υπέρ.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 κατά. Αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 43. Λήξη. Quarante-quatre. Λοιπόν, 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47, 48, 49, 50. Όχι. Καταπίπτουν. Γιατί δεν εγκρίναμε τις 34 και 35. Ε, 53 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά εποχές ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία το όλοι. Λήξη. Απορρίπτεται 16 κατά 12 υπέρ. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 11. Λήξη. Εγκρίνεται 17 υπέρ 11 κατά. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Καταπίπτει. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά εποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά τη 15 λήξη εγκρίνεται 18 υπέρ 11 κατά 16 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 17 υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές να επαληθεύσουμε τη 19. Πέρας εγκρίνεται 19 υπέρ, 11 κατά. 20 υπέρ, κατά. Εποχές, απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά. Εποχές απορρίπτεται, 22 υπέρ, κατά. Εποχές απορρίπτεται, 23 υπέρ, κατά. Εποχές, να επαληθεύσουμε την 23 με ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρχή ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. 17 υπέρ, 12 κατά. 24 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25, 27, 28, 29, 31 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτονται. 26 υπέρ, κατά. Αποχές δεν είναι ξεκάθαρο. Να επαληθεύσουμε για την 26 άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. 16 υπέρ, 14 κατά εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε την 30. Πέρας. Εγκρίνεται 19 υπέρ 10 κατά. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβεστική 1 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το σύνολο της γνωμοδότησης Μονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Μια κάρτα δεν χρησιμοποιείτε. λήξη. Εγκρίνεται 25 υπέρ, 1 5 κατά. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Και ολοκληρώσαμε τις για τα νομοθετικά προγράμματα. Τώρα, θα περάσουμε στην έκθεση Γκάιερ. για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για το Άσυλο. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές, να επαληθεύσουμε τη 2. Ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε για την τροπολογία 4 ηλεκτρονικά. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται 16 ψηφί κατά, 15 υπέρ. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Όχι, ναι. Λήξη. Εγκρίνεται. 28 υπέρ, 3 κατά. Συγχαρητήρια στον κύριο Γκάιερ. Περνάμε στο σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού υπαριθμών 6, έκθεση Μουρεσάν. Δεν έχουμε τροπολογίε. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 21 ψήφους υπέρ 2 κατά. Συγχαρητήρια στον Γενικό Εισηγητή. Να και μια διάταξη Ευχαριστώ, στο Συμβούλιο. Λοιπόν, περνάμε στο Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, έκθεση κατά τη Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, Για την 4, υπέρ. Λοιπόν, μην ε, βιαζόμαστε. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μετά μπορούμε να ψηφίσουμε όντω σε μπλοκ για τις τροπολογίες 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 από την Επιτροπή Απασχόλησης. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το σύνολο της έκθεσης όπως ε, τροποποιήθηκε ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 28 υπέρ, 3 ψήφοι κατά. Συγχαρητήρια στην συγκήτρια. Alors nous maintenant sur le budget 2000. Προπολογισμός 2018. Έχουμε πέντε αιτήσεις μεταφορά. Ο κύριος Ζίκουρντ Μουρεσάν θα μας παρουσιάσει και θα του δώσω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αφού δεν έχουμε προϋπολογισμό για το 2019, ας κάνουμε λίγη δουλειά για τον προϋπολογισμό του 2018. Θα ήθελα να ενημερώσω τους πάντες ότι το 18 είναι ο προπολογισμό για τον οποίο δουλεύουμε έως το τέλος του Δεκεμβρίου. Και ίσως να μας πάρει και λίγο παραπάνω χρόνο τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο. Είναι νωρίς να το πούμε αυτή τη στιγμή. Προς το παρόν όμως πρέπει να, ε, να εγκρίνουμε κάποιες μεταφορές, δεν είναι προβληματικές. Εγώ συστήνω να τις υπερψηφίσουμε όλες αυτές τις μεταφοράς και να σας τις παρουσιάσω γρήγορα. Απόφαση 28 επίπτωση της ε, έκθεσης για ε, Diabaz. Με, μεταφέρουμε 30 εκατομμύρια ευρώ από το απόθεμα του EGF στο, στην κύρια γραμμή του EGF. Δεύτερη μεταφορά είναι η απόφαση 30 που ε, ε, μεταφέρει κάποια ποσά από τη διοικητική γραμμή του ορίζοντα 2020 και του ESI, του ETSF, στις, στα επιχειρησιακά, στις υπηρεσιακές γραμμές ε, αυτών των προγραμμάτων και στο AMIF. 5,95 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Τρίτη μεταφορά είναι η απόφαση 32 που προβλέπει να κατανεμηθούν 3,93 εκατομμύρια ευρώ ώστε να υποστηριχθούν τα πληροφορικά συστήματα και να επανεξοπλιστούν αυτά τις, ε, τα συστήματα της Κομισιόν ως συνέπεια του Brexit. Τα πληροφορικά συστήματα όσον αφορά την Τελωνιακή Ένωση πρέπει να ε, επαναδιευθετηθούν, πρέπει να δοκιμαστούν με τα 27 πλέον κράτη-μέλη προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους αντί των 28 μέχρι σήμερα κρατών μελών και γι' αυτό το σκοπό η Κομισιόν χρειάζεται 3,93 εκατομμύρια. Πώς, ε, πώς ε, ε, διαρθρώνονται αυτά, 3 εκατομμύρια για, την, για τον οργανισμό χημικών από τον οργανισμό χημικών. Εγώ προτείνω να υπερψηφίσουμε αυτή τη μεταφορά για να ενισχυθούν τα πληροφορικά μας συστήματα εν του Brexit. Τέταρτη μεταφορά είναι η απόφαση 33 και αυτή η αφορά ε, προκαταβολή για το κτίριο Ζαν Μονέ 2 που κατασκευάζεται στο Λουξεμβούργο. Το κατασκευάζει το κράτος του Λουξεμβούργου και τον Αύγουστο του 2018 η Κομισιόν μας ενημέρωσε για την πρόθεσή της να ε, καταβάλει μια προκαταβολή ε, στο Λουξεμβούργο. 4,6 εκατομμύρια ε, είχαν καταβληθεί στο τέλος του 2017 και τώρα μιλάμε για 39,9 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα επιτρέψουν στην Κομισιόν να προχωρήσει σε αυτή τη δεύτερη προκαταβολή ποσού προς το κράτος του Λουξεμβούργου. 39,9 λοιπόν για αυτήν την προκαταβολή για το κτίριο Ζαν ε, Μονέ. Από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Μιλάμε για ε, δαπάνε μισθοδοσίας, 3,3 εκατομμύρια ευρώ, 33,3 ε, ευρώ, από, χρήματα από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα τελευταία 2,36 ευρώ θα προέλθουν από την αποκεντρωμένη διαχείριση και όλα αυτά τα χρήματα δεν θα χρησιμοποιηθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς και τα τελευταία 2 εκατομμύρια θα προέρχονται από, δύο, ε, από ε, το εξωτερικό προσωπικό των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 39,9 όπως είπα, συστήνω να την υπερψηφίσουμε και αυτή τη μεταφορά και η τελευταία μεταφορά είναι η απόφαση 35 που προτείνει την μεταφορά 45,2 εκατομμύριων ευρώ για τη χρηματοδότηση των μέτρων αποθήκευσης για την σκόνη από βουτυρωμένου γάλακτος. Αυτό το έχουμε συζητήσει και στη διάρκεια της χρονιάς. Οφείλεται ε, στις απώλειες πωλήσεων ε, στον ε, κλάδο αυτών. Η τιμή αγοράς ήταν χαμηλότερη από την ενδεικτική τιμή που προβλέπεται. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε ένα απόθεμα και ε, έτσι λοιπόν τα κονδύλια του προπολογισμού δεν επαρκούσαν και όπως είπα θα μεταφέρουμε τώρα 45,2 εκατομμύρια ευρώ ε, για τις εκαθαρίσεις των λογαριασμών, από εκεί θα προέλθουν δηλαδή αυτά τα χρήματα και 35,7 από την ε, επίλυση διαφορών και τα τελευταία 500.000 ευρώ θα προέρχονται από την ε, γραμμή της ολοκλήρωσης ε, του, ε, του Τμήματος για την Αγροτική Ανάπτυξη, ΕΧΤΑ και ΕΧΤΕ, 45,2 συνολικά λοιπόν και εδώ συστήνω να υπερψηφίσουμε αυτήν την αίτηση μεταφοράς και με αυτό ολοκληρώνω θα δούμε πώς ακόμα θα μας απασχολήσει αυτός ο προϋπολογισμός του 2018. Άλλο, je me Ευχαριστώ. Ισκιώδης παρακαλώ. Μόνικα, έχετε παρατηρήσει. Συμφωνώ με αυτές τις μεταφορές. Έχει έννοια, έτσι αποφεύγουμε τόκους. Χρησιμοποιούμε πόρους που είναι διαθέσιμοι. Έτσι μειώνονται οι τόκοι και έτσι η αιτήσια επιβάρυνση. Είναι απόλυτα σωστές αυτές οι μεταφορές. Α, αυτή ήταν η σκιώδη του προπολισμού 19 όμως. Ενώ συζητάμε τον προπολισμό του 18. Είμαι υπεύθυνη για τα κτίρια, λέει η κυρία Χολμάη. Εκτό μικροφώνου βέβαια, αλλά ακούγεται. Α, πολύ ωραίο, λέει πρόεδρο. Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Αλλά σας απεκάλεσα ε, σκιώδη για το 19. Για το 18 εννοείστε το 19 καλύτερα. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Κανείς. Ωραία. Να παρατηρήσω ότι εδώ είχαμε προβλέψει υπερβολικά ποσά. Γιατί βλέπω ότι μας περισσεύουν 40 σχεδόν εκατομμύρια, 39,9 και κάτι για την ε, πολιτική ακινήτων. Άρα, κατά πόσο ήταν σωστός ο αρχικός προπολογισμός. Λοιπόν, να τις ψηφίσουμε για τις πέντε μεταφορές από κοινού, αν δεν έχετε αντίρρηση. Ηλεκτρονικά. Άρχεται. Για τις πέντε μεταφορές που μας παρουσίασε ο Γενικός Συγητής. Ψηφίσατε όλοι μου. Ε, ας πούμε, ψηφίσανε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνονται 24 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, μία αποχή. Συγχαίρουμε τον Ζίγκφριντ Μιούρεσαν. Άλλα τμήματα. Και πάλι ο εισηγητής μας. <coughs> Thank you, Chairman. I've got one modification. I've ναι. Έχω πέντε αιτήματα μεταφορών. Τα δύο θα χρειαστεί να ψηφιστούν. Να ψηφίσουμε αφού θα εξηγήσω την ε, φύση των μεταφορών. Πρώτο θέμα. Ελεκτικό συνέδριο. Θέλουν πέντε θέσεις, ε, μόνιμες θέσεις AD να γίνουν ε, προσωρινές θέσεις AD. Έτσι θα μπορέσουν να δώσουν ε, συμβόλαια όριστη ε, διάρκεια για ορισμένους εμπειρογνώμονε που έχουν ήδη επιτόπου. Το στηρίζω. Δεύτερο, ε, επόπτης προστασίας δεδομένων της Ένωσης. Θα θυμάστε ότι ο επόπτης πρέπει να δημιουργήσει ένα ε, σώμα επιτήρησης. Ναι, μεν ε, ίσως να φαίνονται πολλά, 420.000 ευρώ για ένα τόσο μικρό θεσμικό όργανο, αλλά θέλει να δημιουργήσει μια νέα επιτροπή, ένα νέο όργανο για την προστασία των δεδομένων. Ιδιαίτερα θέλουν να ενισχύσουν διάφορες ομάδες, ιδιαίτερα προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για να δημιουργηθεί αυτή η επιτροπή. Δεν χρειάζεται ψηφοφορία από αυτού. Και συμφωνώ με το αίτημα αυτό. Τρίτον, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εξοικονομούν 575.000 ευρώ κατά τη διάρκεια του έτους και προτείνουν να τροφοποιήσουν για να βελτιώσουν την ασφάλεια του κτηρίου τους και να κάνουν και κάποιες επισκευές. Εδώ χρειάζεται ψηφοφορία. Και συστήνω να το εγκρίνουμε. Τέταρτον, Επιτροπή Περιφερειών θέλουν 168.000 ευρώ να μεταφερθούν προς τις εξής τρεις περιοχές. Πρέπει να πληρώσουν για ε, ιδιωτικοποιημένη ε, πληροφορική, θέλουν να φτιάξουν ένα αρχείο για το ίντερνετ τους και θέλουν να κάνουν και κάποιες επισκευές σε κάποια κτίρια. Και τα βρήκαν αυτά τα λεφτά από μειώσεις προσωπικού και από μειώσεις της συντάξης. Δεν χρειάζεται ψηφοφορία. Το στηρίζω. Τέλος. Το Κοινοβούλιο. Δύο αιτήματα μεταφοράς. Πιστώσεων. Πρώτον, C9. Πόροι που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανακαίνιση του PHS και το κτίριο Virts και μια νέα αίθουσα επισκεπτών. Θα τα συμβούλια δεν προωθήθηκαν. Τα ποσά που δεν προωθήθηκαν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν για πληροφορική. Ιδιαίτερα για να αγοράσουν ε, νέο υλικό και για καλώδια και για προγράμματα ε, συνεχούς λειτουργίας ε, των εργασιών του Κοινοβουλίου. Και τέλος η C10 θέλει να χρησιμοποιηθούν πόροι που δεν αξιοποιήθηκαν για αμοιβέ για νέο οπτικοακουστικό εξοπλισμό γιατί είναι πεπαλαιωμένος σε ένα βαθμό. Δεν χρειάζεται ψηφοφορία, το στηρίζω. Δύο ψηφοφορίες λοιπόν Πρώτον για την ΕΟΚΕ, την Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή, και δεύτερον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η μεταφορά C9 για ε, προγράμματα πληροφορική. Συστήνω να υπερψηφίσουμε και τα δύο. Ευχαριστούμε τον κύριο Συγητή. Ερωτήσεις υπάρχουν. Θέλει κάποιος το λόγο. Όχι από ό,τι βλέπω. Επομένως, τέσσερις από αυτές ε, τις ε, μεταφορές μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί, αλλά να ψηφίσουμε την απόφαση 1 που αφορά την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Άρχεται η ψηφοφορία. Tout le Ψηφίσατε όλοι. Λήξη. Εγκρίνεται με 23 ψήφους 3 κατά. Και τώρα ψηφίζουμε τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρχη ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Το C9. Ψήφισατε όλοι. Λήξη. 24 υπέρ, 3 κατά. Συγχαρητήρια στον εισηγητή για τα λοιπά τμήματα. Σε ό,τι αφορά τώρα την κτηριακή πολιτική. Εδώ έχουμε δύο project. Έχουμε πρόταση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης που θέλει να αγοράσει ένα κτίριο στην Νότιο Αφρική για την αντιπροσωπεία της Ένωσης και μια πρόταση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο που θέλει να προβεί σε μεγάλα έργα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των κτίριων. Να δώσω το λόγο στην κυρία Χολμάιερ, τη μόνιμη εισηγητριά μας, για να μας παρουσιάσει εν συντομία αυτά τα έργα και ίσως να θέλουν να πάρουν το λόγο και σκιώδεις συζητές και να απαντήσει η Μόνικα σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Βλέπετε ότι όποτε μου δίνετε τη δυνατότητα εγώ το λόγο τον παίρνω. Λοιπόν, για το δικαστήριο είναι μια ε, εξαιρετικά καλά προετοιμασμένη πρόταση αυτή που μας ε, έχει παρουσιάσει το δικαστήριο με πολλές λεπτομέρειες. Μιλάμε για τον, για εξοπλισμό ασφαλείας του κτηρίου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και τα μέτρα αυτά είναι πραγματικά απαραίτητα. Το δικαστήριο συνομίλησε, ήρθε σε επαφές και με εμπειρογνώμονες ε, και υπηρεσίες των κρατών μελών που ασχολούνται με αυτόν με αυτόν τον τομέα ε, έχουν λάβει συμβουλές ώστε να μην φαίνεται, να μην μοιάζει με φρούριο στο μέλλον το δικαστήριο, να παραμείνει προσβάσιμο και φιλικό, ταυτόχρονα όμως να εξασφαλίζεται και η ασφάλεια. Το κόστος ανέρχεται σε 29,1 εκατομμύρια ευρώ και αυτά είναι 1,6 για το 2019, 17 για το 2020, και 8,5 ε, για το 2000, για το 2021. Το δικαστήριο αποφελείται ε, από τον, ε, από τον κανονισμό, τον δημοσιονομικό, γιατί εκεί ορίζεται ότι δεν, υπα, δεν επιτρέπονται πλέον ενδιάμεση χρηματοδότησης, αλλά πρέπει να ληφθούν δάνεια. 1,85 εκατομμύρια ευρώ ε, εξοικονομούνται με αυτόν τον τρόπο που κανονικά θα πήγαιναν σε ενδιάμεσου. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πόσο καλός και αποτελεσματικό είναι αυτός ο νέος ε, προπολογισμό. Επίση, θετικό είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία με το Λουξεμβούργο, διότι το Λουξεμβούργο πραγματικά διευκόλυνε ολόκληρη τη διαδικασία από την οργάνωση, την προετοιμασία, την εκτέλεση των έργων. Θέλω ρητός να ευχαριστήσω το Λουξεμβούργο γιατί πραγματικά ήταν εξαιρετικά χρήσιμη η συμβολή τους για την κατασκευή αυτών των κτίριων. Το επιτόκιο ε, ορίζεται με τέτοιον τρόπο ώστε το δάνειο να αποπληρωθεί εντός 20 ετών. Φυσικά θα γίνει προσπάθεια να αποπληρωθεί και νωρίτερα. Ε, τα επιτόκια ακόμα δεν έχουν καθοριστεί με απόλυτη ακρίβεια, όμως το Europol συν περιθώριο ε, είναι μια εξαιρετική πρόταση που έχουμε στο τραπέζι, γύρω στο 1% ανέρχεται και έτσι και το κόστος πραγματικά ε, είναι περιορισμένο, είναι εύλογο, δεν δημιουργούνται ε, ακραίες καταστάσεις. Ε, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις, το, η συνολική αξία του κτηρίου ανέρχεται σε 31 εκατομμύρια ευρώ και το κόστος ανέρχεται σε έως το τέλος της ε, ε, διάρκειας αποπληρωμής σε περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ. Ελπίζουμε ότι το, το, το δικαστήριο πρέπει να σας πω ότι ε, με μεγάλη επιμέλεια προσέγγισε τη διαδικασία αυτή, έκανε και μια ανάλυση χειρότερου δυνατού σενάριου, ε, αλλά από ό,τι φαίνεται τα πράγματα είναι πιο καλά. Ακόμη δεν, δεν, υπάρχει, δεν φαίνεται να ε, ευωδώνεται αυτό το χειρότερο δυνατό σενάριο, το οποίο επίση όμως έχει ε, συνυπολογιστεί από το δικαστήριο ε, αυτό ε, θα έλεγα να, να, να προχωρήσουμε κατευθείαν στην πληροφορία για αυτό το ένα, διότι τα στοιχεία για την υπόθεση της Νοτιού Αφρικής είναι λίγο διαφορετικά. Για το πρώτο μέρος, δηλαδή για τις εργασίες σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εδώ δεν υπάρχει αντίρρηση. Οι σκιώδεις συζητητές θέλουν το λόγο. Όχι, να ψηφίσουμε λοιπόν. Ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. «23-2». Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια και στην ε, πεποίθησή τη, ε, στην πειθό της. Τώρα, για την ε, Νότια Αφρική. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο? Ναι. Έχει γίνει καλή προετοιμασία. Έχει γίνει και μια αξιολόγηση κοστοποδοτικότητας για να δει το, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αν θα ήταν καλύτερο αν θα ήταν καλύτερη μια ε, μετακόμιση ή μια κατασκευή νέου κτηρίου ή μια ανακαίνιση του υπάρχοντος κτηρίου η μία περίπτωση θα κόστιζε 5,8 εκατομμύρια, 7,9 το η ανακαίνιση. Παρόλα αυτά, ε, γι' αυτό λοιπόν, ε, ε, μάλλον από τις επιλογές που, που είχαμε στη δυνατότητα στις, ε, μπροστά μας, το 7,1 εκατομμύρια είναι για τη μετακόμιση, είναι η πλέον πρόσφορη ε, δυνατότητα η αγορά ενός νέου κτηρίου λοιπόν είναι η θετικότερη επιλογή που έχουμε μπροστά μας. Ε, βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτικής Δράσης ε, δεν παρίσταται αυτή τη στιγμή ε, στην αίθουσα. Ήθελα να τους απευθύνω το εξής ερώτημα. Γενικά βεβαίως διάκειμε θετικά, ούτε θέλω να ασκήσω κάποια κριτική στην ΕΕΔ, όμως υπάρχει εξής κατάσταση. ε, πολύ συχνά έχουμε να κάνουμε με κτίρια τα οποία δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι ιδιοκτήτε τους, όπου γνωρίζουμε απλώς ε, κάποια δικηγορικά γραφεία τα οποία εκπροσωπούν τους ιδιοκτήτε. Είχαμε αυτό, ε, το, αυτή την περίπτωση και στη Μόσχα. Εκεί θέλαμε πραγματικά να μάθουμε ποιος, ποιος, ποιοι, ποιοι είναι οι δικαιούχοι ε, ποιοι έχουν την κυριότητα του κτίριου. Όχι μόνο ποιοι εκπροσωπούν, που είναι κάποιο δικηγορικό γραφείο, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ε, θέλουμε να ξέρουμε ποιοι είναι οι, ε, οι ιδιοκτήτες, οι πραγματικοί. Εγώ και ο κύριος Κταρό ε, κάναμε μια έρευνα, προσπαθήσαμε να μάθουμε ποιοι είναι τελικά οι ιδιοκτήτε, σε ποιους πηγαίνουν τα χρήματα. Γιατί με βάση το νέο, τη νέα οδηγία για το ξέπλυσμα βρώμικου χρήματο, ε, μας υποχρεώνει να γνωρίζουμε ε, ονομαστικά αν οι ιδιοκτήτε στους οποίους καταλήγουν τα χρήματα ε, είναι επιλέξιμοι, έχουν δικαίωμα. Ε, και αυτό αφορά και εκείνες περιπτώσεις όπου έχουμε νομικά πρόσωπα που βρίσκονται στο προσκήνιο. Ε, στην ε, Νότια Αφρική πάλι έχουμε μια τέτοια περίπτωση λοιπόν. Ε, ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παρεμπιπτόντως. Δεν έχει έρθει ακόμα η ΕΕΔ. Δεν είναι το, το, το, το κτίριο αυτό δεν θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε ξανά στις 10 Δεκεμβρίου. Απλά θέλουμε να μας δώσουν αυτή την πληροφορία αν γίνεται, σε ποιον ανήκουν αυτά τα κτίρια ε, για να μην γνωρίζουμε απλώς ε, το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τον ιδιοκτήτη. Ε, και νομίζω ότι πρέπει και στις δύο περιπτώσεις, και στην Νότια Αφρική και στην Μόσχα, να μάθουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των κτηρίων. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβλημα, εντάξει, να, το ξαναδούμε. Δεν είναι τόσο μεγάλο το, το πρόβλημα. επί του περιεχομένου δεν έχω ανησυχίες, απλά θέλω να μάθω αυτή την πληροφορία και αφορά αυτή η επιθυμία μου τα κτίρια και στη Μόσχα και στην ε, Νότια Αφρική γιατί μαθαίνω ε, όλο και περισσότερο βλέπω ότι έχουμε να κάνουμε με διευθυντές δικηγορικών γραφείων. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω, συμφωνείτε με αυτή, την, ε, με αυτή τη διαδικασία, με αυτή τη μεθοδολογία. Δεν ξέρω, τώρα δεν είναι εδώ και η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Θέλετε να τους περιμένουμε ή θέλετε να μεταφέρουμε το, το, την ψηφοφορία στην συνεδρίαση της 10 Δεκεμβρίου. Ε, μπορούμε να αναβάλουμε, χωρίς πρόβλημα. Ε, μήπως υπάρχουν ερωτήσεις ε, προς την συγκέντρια. Εγώ θα είχα μία. Ξέρουμε ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, ανοίγει όλο και περισσότερα γραφεία ε, σαν πρεσβείες. Μήπως τελικά θα έχουμε 29 πρεσβείες σε κάθε πρωτεύουσα. Μήπως θα μπορούσαμε κάπως να ε, συνδυάσουμε αυτές τις εκπροσωπήσεις μας ε, εκτός Ένωσης για να γλιτώσουμε κάποια λεφτά. Είναι τρομερό αυτό. Ενώ δεν έχουμε εξωτερική πολιτική, να έχουμε τόσες εκπροσωπήσεις. Γιατί κάθε κράτος μέρος έχει κρατήσει τη δική του εξωτερική πολιτική. Νομίζω ότι ξοδεύουμε πολλά λεφτά για κάτι που δεν είναι καθόλου σαφές. Αν αύριο ενώπιον ε, των εκλογέων ε, τεθούν ερωτήματα, εγώ νομίζω ότι θα ζοριστούμε. Ναι, θα απαντήσω ε, με δύο πλευρές στην επιχειρηματολογία μου. Κάπου που υπάρχουν μεγάλα κτίρια, κάποια μικρότερα κράτη-μέλη μπορούν να μπουν σε αυτά τα κτίρια. Αλλά όπου έχω ρωτήσει για τα πέντε μεγάλα κράτη ε, υπάρχει πολλή επιφλακτικότητα να είναι στο ίδιο κτίριο με μια ευρωπαϊκή εκπροσώπηση. Γιατί έχουν και πολλούς συνεργάτες οι μεγάλες αυτές πρεσβείες και τα κτίρια δεν επαρκούν. Θα πρέπει να φτιάξουμε ουρανοξύστες για να έχουν όλοι γραφείο. για την Νότια Αφρική δεν έχει ε, πολύ έννοια αυτό, αλλά θα έχουμε την Τράπεζα Επενδύσεων. Θα είναι υπενικιαστή στο κτίριό μας. Και σε ορισμένες χώρες κάποια κράτη-μέλη που έχουν μικρές πρεσβείες και αυτοί ευχαρίστως ε, παίρνουν κάποια γραφεία στα κτίρια της δικής μας εκπροσώπησης γιατί έτσι λύνουν κάποια θέματα και κόστους, έχουν κοινή πληροφορική, κοινή καλωδίωση, αλλά στις μεγάλες χώρες στην Αμερική και τέτοια, ιδιαίτερα τα μεγάλα κράτη-μέλη το απορρίπτουν. Γιατί εκεί έχουν μεγάλες πρεσβείες. Γιατί δεν χωράνε. Αλλά επίσης ε, γιατί δεν θεωρούν ε, για λόγους προβολής ε, του κράτους τους ότι είναι δυνατόν ένα τέτοιο κτίριο με την ευρωπαϊκή εκπροσώπηση. Αλλά σε κάποιες χώρες υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Σε αυτή την περίπτωση το κτίριο αυτό είναι πολύ κοντά στις πρεσβείες της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, νομίζω και του Βελγίου. Γύρω-γύρω μόνο πρεσβείες έχει. Αλλά η πρόθεσή σας είναι ευγενής κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος. Από ό,τι άκουσα ε, έρχονται οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και επειδή έχουμε χρόνο μπορούμε να διακόψουμε ενδεχομένω ε, δύο λεπτά για να μας δώσουν τις απαντήσεις οι εκπρόσωποι της ε, ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ωραία να διακόψουμε λίγο. Αλλά μην πάτε μακριά. Θα ξαναρχίσουμε πολύ σύντομα. Bien, la séance est reprise. Ωραία, ωραία, επανερχόμεθα. Ε, μην ζητήσετε συγγνώμη, κύριε εκπρόσωποι τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, κυρίε και κύριοι ε, τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Εμεί ε, ε, ήμασταν. Ε, είχαμε ολοκληρώσει λίγο πιο σύντομα τα προηγούμενα θέματα. Η κυρία Χολμάιερ, η εισηγήτριά μας, θα σας κάνει μερικές ερωτήσεις για να διευκρινιστούν οποιασδήποτε, να διασκεδαστούν οποιασδήποτε αμφιβολίες. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη από την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, γιατί κατ' εξαίρεση εμείς ήμασταν πιο γρήγοροι σήμερα, συνήθως είστε εσείς. Είχα τηλεφωνήσει στην υπηρεσία σήμερα ε, και τους ξαναέθεσα το θέμα. Με, βάση την οδηγία για την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων προβλέπεται ότι δεν αρκεί να γνωρίζουμε μόνο τους νόμιμους ιδιοκτήτες, δικηγορικά γραφεία ή οποιαδήποτε εταιρεία που έχει συσταθεί και στην οποία ανήκουν τα κτίρια, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε πραγματικά εκείνου στου οποίου πηγαίνουν τα χρήματα, ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτε των κτίριων. Κατά τα άλλα, ε, συνεχάριν την ε, ε, Υπηρεσία εξωτερική δράση για την επιλογή του κτηρίου, για την προετοιμασία του φακέλου. Δεν έχουμε ανησυχία επί της ουσία, όμως πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των κτηρίων στη Μόσχα και στην Πρετόρια. Ποιοι κρύβονται ή βρίσκονται, εν πάση περιπτώσει, πίσω από αυτές τις δικηγορικέ εταιρείε με τις οποίες ερχόμαστε σε επαφή. Αυτή είναι η ερώτηση μου. Bien. Bienvenue. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών για να μας δώσετε κάποιες διευκρινήσεις. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Είναι σημαντικές ερωτήσεις που ήδη αναφέρθηκαν κατά τον ε, πρώτο φάκελο, όταν μιλούσαμε για την αντιπροσωπεία μας ε, στην ε, Ρωσία, το σημειώσαμε και πολύ πρόσφατα, πριν λίγα λεπτά, στείλαμε κάποιες συμπληρωματικές πληροφορίες στην κυρία Χολμάγερ και είχαμε ένα πρώτο επίπεδο πληροφοριών για τα ονόματα που βρίσκονται πίσω από αυτή την νομική οντότητα Πρόκειται για οκτώ τη της Αφρικής ε, που είναι πίσω από αυτή τη νομική οντότητα. Φυσικά θα προχωρήσουμε και σε πρόσθετη επαλήθευση. Ε, θα πάρουμε αποσπάσματα πρόσθετα από τα Μητρώα και ήδη έχουμε συμπεριλάβει τις νέες διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού και ακριβώς την ενίσχυση επί των άρθρων αυτών. Νομίζω ότι αυτό δεν αφορά μόνο το θέμα της νομοποίησης παράνομων εισόδων, αλλά και θέματα φορολόγησης, γιατί προφανώς μας ε, ενδιαφέρουν και μας ανησυχούν πολύ αυτά τα θέματα. Από τη μία ε, δίνουμε ουσιαστικά παράτρωση στα κράτη να βελτιώσουν τις ε, οικονομικές τους επιδόσεις ε, από τη μια, από την άλλη, ε, ουσιαστικά θα πρέπει να προβαίνουμε και στους κατάλληλους ελέγχους για τη Ρωσία. Εκπλήσωμαι που ξανάρχεται το θέμα. Γιατί νομίζω ότι οι πληροφορίες ε, για τους ιδιοκτήτες, για τα φυσικά πρόσωπα που κρύβονται πίσω από την εταιρεία είχαν σταλεί. Αλλά αν θέλει η Επιτροπή, φυσικά θα το ξανασυζητήσουμε την κυρία Ελχόλμαϊερ, βέβαια για την Νότια Αφρική εμείς ε, έχουμε πάρει και θα αποκτήσουμε και νέες πληροφορίες και θα παρακολουθήσουμε αυτό το ζήτημα. Από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης όμως έχω εφησυχαστεί, γιατί αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να προχωρήσουμε. Η ιδέα είναι ίσως να μην υπογράψουμε απαραίτητα μέχρι τα τέλη του έτου. Αν χρειαστεί, μπορούμε να υπογράψουμε και στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Ε, δηλαδή, δεν έχουμε υποχρέωση, απλώ κινδυνεύουμε να χάσουμε την ευκαιρία γιατί έχουμε και ανταγωνιστεί την πρεσβεία της Κορέας και θέλει αυτό το συγκεκριμένο ε, κτίριο. Όμως, ε, αν περνούσαμε από τη Δημοσιονομική Αρχή, θα μπορούσαμε να ξεκαθαρίσουμε και τις νομικές πτυχές και να αποσαφηνίσουμε και την πρόθεση. Το ερώτημά μου είναι το εξής και το έχω θέσει πολλές φορές. Δεν με ε, απασχολεί σε ποιον ανήκει το δικηγορικό γραφείο. Με ενδιαφέρει να μάθω ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες του κτηρίου. Δεν έχω λάβει αυτή την πληροφορία για, την, ε, για τη Μόσχα. Αν μου τις δώσετε μπορώ να τις διαβιβάσω και στον συνάδελφο Τανά, το ίδιο και για την Πρετόρια. Αφού το κάνετε μπορούμε να εγκρίνουμε και το κτίριο αυτό. Αλλά τις χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες γιατί ε, εμείς ως πληροφορία έχουμε λάβει μόνο τον, ε, τον επικεφαλής, τον ιδιοκτήτη του δικηγορικού γραφείου. Δεν μας ενδιαφέρει όμως, θέλουμε να ξέρουμε σε ποιο θα πάνε τα χρήματα. Γιατί θυμάμαι και τα έγγραφα του Παναμά, όπου ένα καταπληκτικό δικηγορικό γραφείο ε, διαχειριζόταν δισεκατομμύρια ευρώ από μαύρα ταμεία, από φοροδιαφυγή και που στη συνέχεια ε, κατευθύνονταν ε, μέσω ε, ετηριών θηρίδων σε διάφορα ακίνητα και χρειάστηκε να ξετυλιχτεί το κουβάρι μέχρι να, και να γίνουν μεγάλες προσπάθειες μέχρι να μάθουμε ποιοι ήταν τελικά πίσω από όλα αυτά. Γι' αυτό και για εμάς το ζήτημα των ποινικών ευθυνών είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, όσον αφορά τα κτίρια, το, τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Δεν με, δεν με ενδιαφέρει να μάθω ποιος είναι ο πρόεδρος ή ιδιοκτήτης του δικηγορικού γραφείου. Όταν θα λάβουμε αυτές τις πληροφορίες, με χαρά να εγκρίνουμε βεβαίως ε, την πρόθεσή σας αυτή για, την, ε, για το κτίριο αυτό, διότι μας ενδιαφέρει και μας βεβαίως η στέγασή σας. Vous το σύστημα που περιγράφεται είναι ουσιαστικά οι ρωσικές μπάμπουσκες. Ναι, λέει η κυρία Χολμάγερ. Ακριβώς αυτό είναι. Καλούμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να είναι ιδιαίτερα προσεκτική τι καταγγέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους φορολογικού παραδείσους. Δεν μας αρέσουν οι φορολογικοί παράδοσοι στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν φορολογικοί παράδοσοι στην Ευρώπη άλλωστε. Δεν υπάρχει. Ils Νόμιμοι. Αλλά ξέρετε πότε τι γίνεται. Μερικοί είναι πιο νόμιμοι από άλλους. Δεν θα πρέπει λοιπόν να είμαστε καχύποπτοι. Ε, θα πρέπει να, να συμμετέχουμε σε τέτοιες δραστηριότητες που επιτρέπουν την ομοποίηση παράνομων εισόδων. Θα ήταν παράδοξο. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταπολεμήσει όλους τους φορολογικούς παραδείσους ε, και θα πλουστεύσουμε και τη φορολογική μας διαδικασία γιατί η υπερβολική φορολόγηση οδηγεί σε διαδικασίες φορολογικής βαλιστοποίησης. Ε, και Ξέρετε, οι Ευρωπαίοι κάνουν ό,τι μπορούν για να πληρώνουν φόρου. Λοιπόν, έχω μία ακόμη ερώτηση στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ποια είναι η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως ε, θα πρέπει να υπάρχουν τόσες ε, πρεσβείες για να, για να υπάρχει εξωτερική πολιτική. Όμως με ανησυχεί κάπως ε, ότι έχουμε 29 πρεσβείες, 28 αύριο γιατί θα αποχωρήσει η Μεγάλη Βρετανία. Όμως ε, μήπως ε, θα μπορούσε να γίνει σημαντική εξοικονόμηση πόρων, γιατί όταν μιλάμε για μείωση των δημοσίων δαπανών, ίσως ε, από τη σκοπιά της καγκελαρίας μπορούν να γίνουν κάποιες προσπάθειες. Μπορείτε να μας πείτε, πάντοτε έτσι ήταν, πάντοτε χρησιμοποιούσαμε αυτούς τους πόρους, αλλά αν οι συμπολίτε μας το γνώρισαν αυτό, πιστεύω ότι θα το δέχονταν ως έχει. Και αν είχαμε και εξωτερική πολιτική ακούμε πάντα ποια είναι αυτή η εξωτερική πολιτική. Όταν λοιπόν όταν θα έχουμε αυτά τα κτίρια στην Νότιο Αφρική, θα μπορούσαμε να νοικοκυρέψουμε και το τι γίνεται στις καγκελερίες των διάφορων κρατών. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Αλλά κατά την αντιλεγή απόψεων ε, για την κεντρική πολιτική τον Ιούλιο, ήδη είχαμε αναφερθεί σε αυτό το θέμα Προφανώς ε, κατανοείται ότι δεν εξαρτώνται όλα από την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, ούτε καν από τα θεσμικά όργανα και η βούληση των κρατών μελών θα πρέπει να πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση. Όμως, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των ε, υποδομών, εμείς συστηματικά ε, προωθούμε τη συγκατοίκηση και ζητούμε συνέργειες με τα κράτη-μέλη συστηματικά προς αυτή την κατεύθυνση. Στην ε, περίπτωση της Νοτιοαφρικής, ε, ε, δυστυχώς το μέγεθος δεν θα μας επιτρέψει να υποδεκτούμε πολύ περισσότερους. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει προβλεφθεί να συσταγαστεί μαζί μας, αλλά σε μια χώρα όπως η Νότια Αφρική, με τόσο σημαντικό όγκο πρεσβειών, θα ήταν δύσκολο να έχουμε όλα τα κράτη-μέλη μαζί. Έχουμε συγκεκριμένε περιπτώσει όπου λειτουργεί καλά η κατάσταση στην Κάνα, παραδείγματο χάρη, με του Γερμανού από κοινού ε, κατασκευάζουμε ένα κτίριο για να εγκαταστήσουμε τις πρεσβείες. Ε, έτσι λοιπόν μπορεί να γίνει εξοικονόμηση πόρων και οι Υπουργοί Οικονομικών θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν περισσότερο παρά οι Υπουργοί Εξωτερικών γιατί ίσως ο καθένας ε, θα θέλει να διατηρήσει τη δική του ζώνη επιρροής και δεν βλέπουν απαραίτητα καλό να είναι όλοι υπό την ίδια στέγη. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό στην Τανζανία σε ένα κτίριο όπου Εμεί συστεγάζονται, Εμείς από την πλευρά μας προωθούμε αυτές τις προσπάθειες, τυποποιούμε τα έγγραφα για να το διευκολύνουμε αυτό. Έχουμε τριπλασιάσει τον ε, αριθμό των συστεγάσεων τα τελευταία τρία έτη. Γίνεται δηλαδή κάτι συχνό και έχουμε μια ειδική ομάδα ε, που ασχολείται με αυτό το θέμα και στο μέτρο του δυνατού προσπαθούμε να το προκαλέσουμε προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή να υποδεχτούμε τα κρατημέλη ή εμείς να συστεγαστούμε στα κτίρια άλλων κρατών μελών. Συμπληρωματική ερώτηση στην Νότιο Αφρική. Πόσες πρεσβείες ε, έχετε εντοπίσει που εκπροσωπούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ε, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Πάνω από 20, αλλά σίγουρα όχι όλα τα κράτη-μέλη. Δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη χωριστέ πρεσβείε, αλλά ίσω 21-22. Δυστυχώ δεν την έχω αυτή την τροφόρηση. Αλλά είναι μια χώρα όπου υπάρχει εκτεταμένη εκπροσώπηση των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ ο πρόεδρο. Ωραία. Εντάξει, αρκεί κυρία εισηγήτρια. Έχετε άλλε ερωτήσει, Ευχαριστώ πολύ. Α, ε, ναι. Ναι. Θέλω να πω ότι μόλις μας δώσετε τα αναγκαία έγγραφα θα εγκρίνουμε. Θα εγκρίνουμε αμέσως για να αποφύγετε να σας το πάρει η Κορέα. Μόλις μας δώσετε την κατάλληλη προφόρηση θα, που θα μπορούσα να στείλω στου σκιώδει, θα εγκρίνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, η μόνη ε, ημερομηνία που μας μένει λοιπόν είναι 10 Δεκεμβρίου, μέχρι τότε έχουμε τα, τη, την αναγκαία πληροφόρηση. Για την περαιτέρω πολιτική κτηρίων έχετε άλλα θέματα κυρία εισηγήτρια, όχι. Ωραία. Οπότε, να περάσουμε τώρα. έλεγχος των συνόρων. Ευρωπαϊκή άκτο και φυλακή. Γιάννης Γκάια να παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης και κατόπιν οι εφόσον θέλουν να εκφραστούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι. Μιλάμε για τον οργανισμό με το όνομα Frontex, που είναι γνωστό τώρα σε όλους, που πλέον ε, μετονομάζεται σε ακτοφυλακή και συνοριοφυλακή και θα ε, χρειαστεί να συνηθίσουμε το, αγγλικό αρκτικό αλεξοβή BCGA. Μιλάμε στην ουσία για τη Frontex. στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2019 έχουμε κάνει ήδη το νέο, το πρώτο βήμα για αυτόν τον οργανισμό. Έως το 2020 ο οργανισμός αυτός θα έχει, ένα, θα έχει προσωπικό 10.000 ατόμων, εκ των οποίων οι 3.000 θα ανήκουν στον οργανισμό, 3.000 ε, θα είναι αποσπασμένοι των κρατών μελών και ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να ε, προσλαμβάνει με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ε, εμπειρογρόμονες και αξιωματούχους από τα κράτη-μέλη. 4.000. Πρόκειται για γιγάντιο έργο και για να προχωρήσουμε με έφτακτο τρόπο έχουν ήδη προσημειωθεί 20 ε, εκατομμύρια για τον οργανισμό, 375, 375 ε, θέσεις απασχόλησης, δεν υπήρξαν ε, και διαφωνίες και ο συνολικός προπολογισμός αυτού του οργανισμού θα ανέλθει για την συνολική περίοδο του πλαισίου σε 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Επειδή η, ατομική, η Επιτροπή Ατομικών Ελευθεριών έχει προβλέψει και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον κανονισμό, ε, εγώ περιορίστηκα σε συγκεκριμένα θέματα. Σε αυτά συγκαταλέγονται η επανάληψη της θέσης του Κοινοβουλίου του 2016 ότι εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε αρμοδιότητα στον οργανισμό αυτό να παρεμβαίνει και σε τρίτες χώρες όσον αφορά την ε, επιστροφή ε, επιστρεφωμένων προσώπων. Ε, το συζήτησα και με τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού αυτό σήμερα. Συμφωνούμε σε αυτό. Σε πρώτη φάση ο οργανισμός να δραστηριοποιηθεί στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και αρκετά φιλόδοξη ήδη αυτός ο στόχος προτού αναθέσουμε στον οργανισμό και καθήκοντα στο εξωτερικό, σε τρίτες χώρες. Θα πρότεινα επίσης να ενισχύσουμε τον εποπτικό ρόλο του Κοινοβουλίου και να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και ξεκαθαρίζουμε ότι κατά την ε, κατάρτιση του πολιετούς ε, προγράμματος εργασιών ο οργανισμός θα πρέπει να λογοδοτεί και στο Κοινοβούλιο να λαμβάνει υπόψη του την εξοικονόμηση πόρων και να λάβει υπόψη του την σύσταση ε, του, της ε, διοργανικής ομάδας εργασίας πέρσι για τον βασικό κανονισμό. Ε, μία αλλαγή επίσης θέλω να απαλληφθεί. Δεν θέλουμε να δοθεί ε, ε, η υποχρέωση, ή ε, μάλλον η δυνατότητα ο οργανισμός να λαμβάνει μεταφράσεις και στην ελεύθερη αγορά. Υπάρχει ε, υπηρεσία στο Λουξεμβούργο, σχετική και αρμόδια, εξειδικευμένη και η Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού, του, της υπηρεσίας μάλλον, μου ζήτησε να μην δοθεί μια τέτοια δυνατότητα στον οργανισμό, στην Frontex, διότι τα προβλήματα έχουν ξεπεραστεί, πλέον είναι λειτουργική η υπηρεσία και ε, διότι η υπηρεσία αυτή δεν θα μπορούσε να συνεχίσει το έργο της αν επιτρέπεται σε άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς να απευθύνονται για τις μεταφράσεις τους στην ελεύθερη αγορά. Ε, προτού ε, βεβαίως οι χριστιανοδημοκράτες μου πούν ότι επιτίθαμε στην ελεύθερη αγορά, θα σας πω ότι το 90% ε, των, ε, ε, των μεταφράσεων της υπηρεσίας αυτής προέρχονται από την ελεύθερη αγορά Απλώς ε, εκεί όπου υπάρχουν ειδικέ απαιτήσει ε, ασφάλειας ή ποιότητας ε, κάνει εσωτερικά τις μεταφράσεις της. Οπότε νομίζω ότι η ποιοτητα κανει εσωτερικα τι μεταφρασει αυτή θα ήταν έολη αν μου απευθυνόταν. Ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση. Για αυτήν την τόσο σημαντική πρόταση για ένα θέμα που είναι στο επίκεντρο των ανησυχιών μας. Είναι ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Επ' αυτού Θέλει κανένα το λόγο. Ο κύριος ε, Σάρβαμα. Ευχαριστώ κύριε Γκάιερ για το σχέδιο γνωμοδότησης. Φυσικά συμφωνώ ότι χρειάζεται περισσότερο συντονισμός ε, όσον αφορά τη, τα καθήκοντα εξωτερικών και άμυνα σε τρίτες χώρες. Είμαι και υπέρ των τροπολογιών σας 5 και 6 για να βελτιωθεί η διακυβέρνηση αυτού του οργανισμού. Ωστόσο, διαφωνώ με τις τροπολογίες σα 1, 2 και 3. Κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντικό ο οργανισμός αυτός να είναι σε θέση να λειτουργεί και να στηρίζει τρίτες χώρες για τις επιστροφές. Καταλαβαίνω τα επιχειρήματα. Ότι πρώτα να αρχίσει να λειτουργεί αυτός ο οργανισμός τουλάχιστον στη δική μα επικράτεια αλλά αυτό είναι ένα θέμα παγκόσμιο, δεν σταματάει σε σύνορα. Η αποτελεσματικότητα, η... όλος ο λόγος ύπαρξης ε, ενα... ενός τέτοιου οργανισμού εάν δεν μπορεί υπαρξης ενό ενος τετοιου οργανισμου εαν δεν μπορει ευθυ εξ αρχή ε, να λειτουργεί παντού στον κόσμο, εκτό των συνόρων δηλαδή, τότε θα ήταν ε, λυψό. Θα έπρεπε από την αρχή να έχει αυτή τη δυνατότητα και έτσι θα προσέφερε και ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Για την αποτελεσματικότητα και τα αποτελέσματα νομίζω ότι αυτό το σώμα των 10.000 θα πρέπει κυρίως να αποτελείται από σπασμένους από τα κράτη-μέλη με μακροχρόνιες αποσπάσεις. Οπότε τα κράτη-μέλη θα είχαν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι αυτό το σώμα δημιουργείται, αυτό το μόνιμο σώμα λειτουργεί και είναι λειτουργικό Επίσης, η υπεραιτέρω ε, ενίσχυση αυτού του οργανισμού δεν θα πρέπει να δημιουργήσει επικαλύψεις με τη λειτουργία των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, θέλει σα το λόγο. Δεν βλέπω. Το θέμα που ανέφερε ο κύριος Σαρβαμά είναι ζωτική σημασία. Θα σταματάμε στα σύνορα τρίκτο σένσου ή θα προσπαθήσουμε να σταματήσουμε τις μεταναστευτικές ροές πιο, πιο μπροστά ακόμη, δηλαδή και στις χώρες μετάβασης. Στη Λιβύη, για παράδειγμα. Αν διαπιστώσουμε ότι κάπου δεν λειτουργούν τα κράτη, τα κράτη ε, από τα οποία περνάνε οι μετανάστες και επειδή δεν υπάρχει κράτος ε, διάφορες εγκληματικές ομάδες οργανώνουν και προωθούν τις μεταναστευτικές ροές. Αυτό βέβαια θα προκαλέσει πολύ έντονες συζητήσεις. Κύριε Γκάιερ, για να ολοκληρώσετε. Ναι, πράγματι. Ε, διαφωνώ. Έχω μια διαφορετική οπτική. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ο νέος οργανισμός να λειτουργεί εντός ενός νομικού πλαισίου μέσω του οποίου εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι δραστηριότητες αυτού του οργανισμού θα ε, εκτελούνται υπό την τήρηση της νομιμότητας και των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για τις τρίτες χώρες ε, και εκείνες που αναφέρετε εσείς, δεν νομίζω ότι μπορεί αυτό να εξασφαλιστεί. Ποιος μας λέει ότι μια επιστροφή από τη Λιβύη ε, ε πραγματοποιείται νομίμως και ότι οι άνθρωποι που επιστρέφονται από τη Λιβύη στις χώρες καταγωγής τους ε, γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματά τους. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να προχωρήσουμε σε έναν πιο εξειδικευμένο ορισμό ε, στις, ε, για υποψήφιες χώρες, από τις οποίες, για παράδειγμα, αναμένουμε ότι θα τηρούν το νομικό πλαίσιο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί έχω μιλήσει και με τον Γενικό Διευθυντή ε, και είχαμε την ιδέα ότι θα μπορούσαν ενδεχομένω να, να, να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό άλλων χωρών. Παραμένω στο παράδειγμά σα, να βοηθήσουμε για παράδειγμα την Λιβύη, οι αστυνομικέ, τελωνιακέ, συνοριακέ αρχέ, όποιο και αν εμπλέκεται σε μια τέτοια διαδικασία, να μπορούν να εκτελούν τι επιχειρήσει του με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όσο πιεστικό και αν είναι το πρόβλημα, το να δώσουμε αυτή τη στιγμή στον οργανισμό την αρμοδιότητα να παρεμβαίνει όπου κρίνεται από ποιον αναγκαίο, ε, νομίζω ότι θα ήταν υπερβολικό σε αυτή τη φάση. Μία συμπληρωματική ερώτηση αν επιτρέπετε. Ναι, οι οργανισμοί, ναι, οι φορ... Μα ο Φράντεξ είναι. Ναι μέχρι τώρα είχε το όνομα Frontex και τώρα παίρνει το όνομα Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Είναι λίγο αυτό το κουραστικό ακρόνιμο EBCGA. Ναι, λέει ο πρόεδρος. Και η έδρα του θα παραμείνει στη Βαρσοβία. Ναι, λέει ο κ. Γκάιερ. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρος. Ωραία. Ωραία, είναι ένα διευρυμένο Frontex. Και μετονομασμένο αλλά είναι πάντα ο οργανισμός Frontex. Ωραία. Δύο συνάδελφοι θέλουν τον λόγο. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν θέλει κανείς τον λόγο. Οι τροπολογίες πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 3 η ώρα της 20 ης Νοεμβρίου, δηλαδή αύριο. Στις 10 Δεκεμβρίου θα ψηφίσουμε Η ΛΥΜΠΕ είναι η επιτουσίας αρμόδια, η οποία θα ψηφίσει στις 23 Ιανουαρίου. Τώρα να περάσουμε. ΕΝΤΕΙΣΕΙ Το μέσο για την ανάπτυξη της γειτονίας και για τη διεθνή συνεργασία. Και η Εντέρ Καρδιαθάβαλ θα μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ παρουσιάζω την γνωμοδότηση πώς η Επιτροπή Προπολογισμών θα πρέπει να στείλουμε στην Επιτροπή Ανάπτυξη και Εξωτερικών Υποθέσεων για αυτό το μέσο Γειτονία ανάπτυξη και διεθνού ε, Συνεργασία. Εντίτσι το λέμε εμεί. Ε, αντί να λέμε όλη αυτή τη φράση. Λοιπόν, η Επιτροπή Δυνάμει του άρθρου 54 είναι αρμόδια για ορισμένα τμήματα. Για να ξέρετε για τι πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για αυτό που θα διαδεκτεί ε, το μέσο του FCD e που έχουμε, που έχουμε διεργαστεί στην Επιτροπή μας. Έχω καταθέσει, έχουν κατατεθεί 59 τροπολογίες, όμως μπορούμε να τις δούμε σε διάφορα μπλοκ. Καταρχήν για τα αριθμητικά στοιχεία όπως ε, κάναμε και για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουμε προσαρμόσει σε ε, σταθερές τιμές ε, όλα τα νούμερα και αποφασίσαμε να προβούμε σε μια αύξηση στο τμήμα που αφορά την Αφρική για 3,5 ε, δισεκατομμύρια γιατί η Αφρική δεν είναι μόνο μία νέα περιοχή αλλά το ένα τμήμα έχει να κάνει με τη γειτονία και ένα άλλο τμήμα της Αφρικής με την υποσαχάρια Αφρική. Έτσι λοιπόν έχουμε κάνει μία αναλογική κατανομή. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη γραμμή που διέπει τροπολογίες. Τώρα δεύτερον μιλάμε για την εγγύηση που πρέπει να δώσει αυτό το μέσο και πόσα χρήματα θα πρέπει να δώσουμε στην εγγύηση αυτή με αυτό το νέο μέσο εξωτερικής πολιτικής. Ε, ουσιαστικά συγχωνεύονται διάφορα εργαλεία, διάφοροι μηχανισμοί που ήταν ξεχωριστοί μέχρι τώρα. Δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς Πώ θα πρέπει να εφοδιάσουμε την εγγύηση. Επομένω, η πρόταση της Επιτροπής είναι το ποσοστό του εφοδιασμού να πηγαίνει από το 9% που ανταποκρίνεται στην προηγούμενη εξωτερική θητεία της ε, Τράπεζας Επενδύσεως ε, μέχρι το 20% που αφορά το EFSD. Δηλαδή μπορούμε να μιλάνουμε από 36 εκατομμύρια και πάνω. Γι' αυτό προτείνω, έχουμε μια πολύ μεγάλη ψαλίδα, να βάλουμε δηλαδή ένα όριο 10 δισεκατομμυρίων σε αυτή τη μόχλευση της εγγύησης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε έναν έλεγχο για το ποια χρήματα θα δεσμευτούν για τη χρηματοδότηση της εγγύησης και επομένως ε, να μην μειώσουμε τα κονδύλια ε, για τις επιχορηγήσεις ε, σε ένα σημαντικό ε, ποσό όπως είναι τα 30 δισεκατομμύρια. Είναι μέτρο ασφαλείας. Αυτό μπορεί να αλλάξει πάντως και αν ε, εκτιμάει η Επιτροπή ότι πρέπει να πάμε παραπέρα, ε, τότε και η Κομισιόν ή το Κοινοβούλιο μπορούν να ζητήσουν τροποποίηση μέσω κατεξουσιοδότησης πράξης και θα μπορεί να γίνει η τροποποίηση αυτή. Τρίτη μεγάλη γραμμή εργασίας σε αυτό το μηχανισμό, η Κομισιόν προτείνει ένα αποθεματικό, ένα στρώμα το αποκαλεί, ένα μαξιλάρι, που απριόρι δεν θα απευθύνει στις πολιτικές. Μιλάμε για 10 δισεκατομμύρια, 200 εκατομμύρια. Προτιμούν να το αφήσουν αυτό κατά μέρος και ανάλογα ε, με τις μελλοντικές συνθήκες ε, και φυσικά αυτό συμβαίνει πάρα πολύ στην εξωτερική πολιτική και στην ε, αναπτυξιακή συνεργασία. Προτιμούν να αφήσουν αυτά τα 10 δισεκατομμύρια χωρίς να έχουν ήδη κατανεμηθεί. Πιστεύω ότι από δημοσιονομική σκοπιά αυτό είναι πολύ λογικό, να μην έχουμε μπλοκάρει ήδη όλους τους πόρους, να μην έχουμε κατανεμεί ήδη όλους τους πόρους, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε κάποιου μηχανισμού ελέγχου για το πώ θα γίνει η κατανομή αυτών των κονδυλίων όταν θα είναι απαραίτητο. Και γι' αυτό εμεί έχουμε καταθέσει τροπολογίε, δηλαδή ότι αυτό το αποθεματικό, αυτό το μαξιλάρι να ενεργοποιηθεί σύμφωνα με τη δημοσιονομική διαδικασία αν ε, γινόταν ταυτόχρονα με τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, αλλά αφού θα έχει γίνει μια συζήτηση για τις πολιτικές προτεραιότητες με την ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Ανάπτυξη, αν πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια του έτους, να γίνει μέσω μιας μεταφοράς και έτσι και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει το πράσινο φω στην ενεργοποίηση αυτού του επιθεματικού. Τέταρτη γραμμή εργασία είναι ότι σε όλο το θέμα της ενημέρωσης. Έχω βάλει το Κοινοβούλιο στο ίδιο επίπεδο με το Συμβούλιο, γιατί πολλές φορές ε, λέει η Επιτροπή θα στείλει ενημέρωση στο Συμβούλιο και έχω βάλει εγώ και στο Κοινοβούλιο, σε κάθε γραμμή που γίνεται αυτή η αναφορά. Και η πέμπτη μεγάλη γραμμή εργασίας, ε, η Κομισιόν, στα παραρτήματα παρουσιάζει τόσο τους πολιτικούς στόχους όπως και τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση του Ταμείου. Είναι πραγματικά όντως ε, τμήμα του κανονισμού το παράρτημα, αλλά όταν μιλάμε για τέτοια θέματα όπως η διακυβέρνηση και η πολιτική στόχοι, νομίζω ότι είναι καλύτερα να μπει στο διατακτικό. Επομένως θέλουμε να βάλουμε τα παρατήματα στο διατακτικό. Και κάτι ακόμα, γιατί φέρθηκα σε πέντε κατά τις γραμμές, αλλά είναι έξι, έχει να κάνει με, ως, με τις για την έκρηση του Ταμείου Βιώσιμης Ανάπτυξης στην διαφάνεια, ε, τον έλεγχο, τον μηχανισμό καταγγελιών και όλο το τμήμα του ελέγχου και της υποβολής εκθέσεων που πρέπει να κάνει η Κομισιόν κατά τη χρήση του Ταμείου, όλα αυτά που πρέπει να υποβάλει στο Κοινοβούλιο. Όλα αυτά τα διαπραγματευτήκαμε πρακτικά λιγότερο από ένα χρόνο πριν και τα έχουμε πάρει από το Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης και τα προτείνουμε σε αυτό το νέο μηχανισμό γειτονίας ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασία. Μία τελευταία ενημέρωση γιατί ενώ προτιμάζα τη γνωμοδότηση εξ ονόματος της Επιτροπής Προπολογισμών, είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τους τέσσερις εισηγητές ε, από την ανάπτυξη και την εξωτερική πολιτική και επί της αρχής συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό. Είχα συνεδριάσεις μαζί τους, τους εξήγησα ποιες, ποιοι είναι οι στόχοι και προσπάθησα να απαντήσω στις αφιβολίες τους σε σχέση με τον έλεγχο από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Συμφωνούν ότι η δημοσιονομική διαδικασία ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με έναν τρόπο έτσι ώστε να έχουμε έλεγχο της χρήσης του Ταμείου και προφανώς ε, ε, υπάρχουν Υπάρχει πολύ μεγάλη συμφωνία με τους τέσσερις συζητητές ε, για το πώς διαχειριστούμε αυτό το τομείο. Απομένει βέβαια να δούμε και τις τροπολογίες των ομάδων. Ευχαριστώ, Άιντερ, για αυτές τις διευκρινήσεις. Σίγουρα πολύ σημαντικό αυτό το μέσο. για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και για να στερεύσουν οι πηγές μετανάστευσης οι πηγές της μετανάστευσης. Ποιος είχε στο λόγο, ο Ρίμπιχ. Ευχαριστώ την Έντερ. Αυτή η αναδιάρθρωση μιας πολιτικής που ήθελε πραγματικά μεγάλη αναθεώρηση και επειδή η αναπτυξιακή πολιτική ε, είναι βασική πολιτική και η επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων όντως θα παίξει μεγάλο ρόλο. Το θέμα αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν ήδη κάποιες δομές. Άρα πρέπει να προσέξουμε να μην δημιουργήσει και άλλες δομές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται αυτές που ήδη υπάρχουν. Και οι υπάρχοντες οργανισμοί να αναπτύξουν περισσότερο τη δυνατότητα δράσης τους διότι αυτοί οι οργανισμοί ούτως ή άλλως δουλεύουν πολύ καλά. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούν καλύτερα οι υπάρχουσες δομές με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Όλα αυτά πρέπει να αναφέρονται ακριβώ σε εκτελεστικέ διατάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Καρδιαθάβαλ, όπως και στη συζήτηση για το Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης, έκανε ε, ε, πολύ καλή δουλειά που μας επιτρέπει να συζητήσουμε αυτό το σχετικά νέο μέσο, ούτως ώστε να ενταχθεί στη δουλειά μας, αυτό το εντίτσι. Θα πρέπει να μάθουμε και αυτό το ακρόνιμο. Σωστό είναι που θέλετε να υπάρχουν αυτές οι ρήτρε διαφύλαξης και ο έλεγχος από το Κοινοβούλιο και οι διατάξει για την διακυβέρνηση αυτού του νέου μέσου. Γιατί η Κομισιόν παρέλειψε ορισμένα στοιχεία που θα έπρεπε να είναι σε αυτό το κείμενο. Συμφωνούμε ιδιαίτερα λοιπόν με τη γραμμή που έχετε πάρει. Ίσως όμως να υποβάλω μερικές πολύ λίγες τροπολογίες. Μία για να τονίσω το ρόλο των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΣΑ και του ΟΗΕ για τη λειτουργία των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μεγάλων πολυεθνικών. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Θέλουμε έναν ε, συγκεντρωτικό μηχανισμό αντιμετώπισης ε, παραπώνων που, όπου να μπορούν να προσφεύγουν όλοι όσοι επηρεάζονται από τη λειτουργία αυτού του ταμείου, εάν δεν είναι ικανοποιημένοι. Εφόσον δεν έχουν ε, ικανοποιηθεί τα αιτήματά τους από τους μηχανισμούς παραπώνων των ε, ε, συμμετεχόντων. Ο στρατιωτικός τομέας και ο τομέας ασφάλειας πρέπει να είναι χωριστός βέβαια. Και επίση τα θέματα των ρηκτών καυσίμων και τη δέσμευση του άνθρακα. Τώρα που καταλαβαίνουμε τη σημασία τη κλιματική αλλαγή, πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αυτά. Ξέρω ότι είχατε πολλέ συζητήσει σήμερα, δεν θέλω να σα επιβαρύνω. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ την συγγήτρια για το εξαιρετικό έργο της. Συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα είπε, ιδίως όσον αφορά τις διαφορές και την σωστή ισορροπία μεταξύ ε, εχέγιων εξασφαλίσεων, χρηματοδοτικών μέσων, ε, την κινητοποίηση των, ε, των αποθεμάτων και πώς μπορούν όλα αυτά να βελτιωθούν στον κανονισμό και συμφωνώ απόλυτα ε, με αυτό που κάνατε να μεταφερθούν, να μεταφερθεί το ζήτημα της διακυβέρνησης ε, ε, από το παράρτημα στο διατακτικό. Η ανησυχία μου αφορά το γεγονός ότι στον κανονισμό, στην πρόταση κανονισμού, έχουμε το EFSD συν ως μια πλήρως ανοιχτή πλατφόρμα για οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Και εδώ ε, σκέφτομαι την συνέχιση των ε, δράσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Καλό είναι να είναι ανοιχτή αυτή η πλατφόρμα, αλλά θα πρέπει να είναι τελείως ανοιχτή ή μήπως θα ήταν καλύτερα ένα τμήμα ε, του Ταμείου να είναι εξειδικευμένο, να, να επικεντρώνονται πιο πολύ στην, στην ΕΤΕΠ, για να μπορεί να συνεχίσει τις δράσεις της στην Αφρική, στην Καραϊβική, Νομίζω ότι αυτό, αυτό είναι μια διαδικασία που πρέπει να συνεχιστεί και να εξασφαλιστεί η συνέχεια της. Όταν κοιτάμε όλα τα χρηματοστατικά δράματα που μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό το νέο ταμείο, το AFD, η Παγκόσμια Τράπεζα και άλλοι, εκείνοι έχουν ήδη συγκεκριμένες δράσεις που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές και ε, το Ταμείο απλά λειτουργεί συμπληρωματικά. Ε, ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως Ευρωπαϊκή Τράπεζα έχει ειδική σχέση και επίσης υπενθυμίζω ότι λογοδοτεί και στο Κοινοβούλιο. Και το γεγονός ότι η ΕΤΕΠ διαχειρίζεται αυτά τα κονδύλια μας δίνει τη δυνατότητα εμείς να επηρεάζουμε τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Και εδώ δεν είναι το ίδιο ε, με το να είναι κανείς μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με το να είναι ε, το σώμα που συμμετέχει στη λήψη απόφασης. Πρέπει νομίζω να το σκεφτούμε ποιο, ποιο κομμάτι του ταμείου πρέπει να είναι ανοιχτό και ευέλικτο και ποιο θα πρέπει να υπάγεται στην ΕΤΕΠ. Λαμβάνοντα υπόψη και την ανάγκη ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το πώ θα εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα να επηρεάζουμε τα πράγματα στην ε, λήψη αποφάσεων και στον τομέα τη πολιτική αλλά και από γεωγραφική σκοπιά. Ξαναδώ το λόγο στην εισηγήτριά μα που νομίζω ότι θα ευχαριστήθηκε από τα σχόλια που άκουσα. Να δώσω το λόγο στη Γενική Διεύθυνση Ντεύκο ο κύριος Σο, διευθυντής, είναι εδώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να εξηγήσω ορισμένα στοιχεία για την πρότασή μας για ένα μέσο για τη γειτονία, την ανάπτυξη και τη διεθνή συνεργασία. Στα γαλλικά το ακρονίμιο είναι επίσης ε, με αρκετά κακό ήχο. Αν σκεφτείτε κανένα καλύτερο ακρονίμιο ή εσείς ή η εσεις η η ε, να μου το προτείνετε γιατί εντύτσι τώρα λέμε τα επόμενα 8 χρόνια και εσείς και εμείς δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, κυρία Καρδιαθάβαλη. ε, θα ήταν πιο απλό να σας μιλήσω ισπανικά. Καταρχάς, σας ευχαριστώ για την έκθεσή σας. Κυρία Καρδιαθάβαλ, αναφερθήκατε σε 5-6 πλευρές ε, της εργασίας σας. Βεβαίως θέλετε να αυξηθεί το τμήμα των πιστώσεων για την εξωτερική δράση. Τώρα δεν χρειάζεστε εμένα για να σας εξηγήσω ε, πώς εντάσσονται τα ποσά που προτείνονται εδώ στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και ιδιαίτερα στην εξωτερική δράση της Ένωσης. Βεβαίως, μια αύξηση θα μας επέτρεπε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Δεύτερον, προβλέπονται λοιπόν ε, χρηματοδοτήσεις μεταξύ 9 και 50% και να ξέρουμε εκ των προτέρων τι ποσό θα είναι επιδοτήσεις για τη βοήθεια για την ανάπτυξη και πόσα θα πηγαίνανε για τις εγγύσεις του EFSD συν. Θεωρούμε ότι πέρα από ένα διαχωρισμό το βασικό είναι να δούμε τι θα γίνει με τον προγραμματισμό, ποιες είναι οι ανάγκες. Τα 60 δις λοιπόν που προτείνονται δεν είναι ε, κάτι που πρέπει να επιτύχουμε, είναι το απόλυτο μέγιστο. Πρέπει να δούμε ποιες είναι διάφορες δυνατότητες. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια κάποια ευελιξία, είναι σημαντική. Και το ποσό που θα πάει για επιδοτήσεις και το ποσό που θα είναι εγγύηση πιστώσεων, αν εγκριθεί η πρόταση της Κομισιόν, όπως έχει τώρα, συνολικά λοιπόν θα άφηναν τις επενδύσεις στο επίπεδο που είναι τώρα. Δεν θα χάνανε δηλαδή τίποτε οι επενδύσεις, απλώς θα είχαν περισσότερα χρήματα για να συνεργαστούμε με τον ιδιωτικό τομέα. Και όπως λέμε πάντα εδώ, για να εργαστούμε, για να κάνει επενδύσεις ο ιδιωτικός τομέας στην βιώσιμη ανάπτυξη. Τώρα για αυτό το σεντούκι, και αυτή τώρα η έκφραση, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλύτερη στα ισπανικά, η πρόταση της Κομισιόν θα προσπαθήσει να αντιδράσει σε όλα τα πρόπτα όπως αυτές που έχουμε τα τελευταία χρόνια και που θεωρούμε ότι θα συνεχιστούν. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί στο ίδιο επίπεδο και η αναπτυξιακή βοήθεια που δίνει η Ένωση. Γιατί είναι υψηλή προστιθέμενη αξία, γιατί είναι προγραμματισμένη, προβλέψιμη, μακροπρόθεσμη. Αλλά βέβαια αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πολύ περιθώριο για να αντιμετωπίσουμε τα απρόπτα. Γι' αυτό προτείνουμε αυτό το σεντούκι. Αυτό το ποσό θα μας επιτρέψει να ε, χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που υπάρχουν και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, που και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο αποθεματικό. Για πρώτη φορά σε 60 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης να καταργηθεί και οι δαπάνες που κάνουμε για τις χώρες της Αφρικής που είναι το σημαντικότερο τμήμα της εξωτερικής μας δράσης μαζί με τα ποσά για, το, την Αφρική, για την καρεβική και τον Ειρηνικό να μπουν όλα στον προπολογισμό και να είναι λοιπόν υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι λοιπόν θα έχουμε μια διαφορετική μέθοδο εργασία που θα βασίζεται στη διαδικασία του προπολογισμού. Αυτός είναι ένας ε, τρόπος, μια μέθοδος εργασίας που θα πρέπει να αξιοποιήσουμε. Βεβαίω, ε, αυτός ο τομέας δίδει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σημαντική δυνατότητα να παρέμβουν, αλλά δεν είχε χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα. Όπω είπε ο κ. Ρούμπιχ, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέε δομέ, πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτές που υπάρχουν για να ενισχύσουμε τον έλεγχο. Για τον ίδιο λόγο, για την ενημέρωση βεβαίω και για τη διακυβέρνηση πρέπει να εργαστούμε και ε, του νέου Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και για το σύνολο της πρότασης. Και υπάρχουν ορισμένα στοιχεία όπου αν συγκρίνουμε την ε, πρόταση που υπάρχει τώρα για το Ταμείο Βιώσιμη Ανάπτυξη ΣΥΝ με την προηγούμενη ε, λειτουργία του Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη φαίνεται ορισμένα στοιχεία να έχουν αφαιρεθεί. Θέλουμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα για να έχουμε λιγότερη νομοθετική εργασία. Τα περισσότερα που λείπουν ή που θα μπορούσαν να λείπουν θα είναι στο νέο, είναι στο νέο δημοσιονομικό κανονισμό, οπότε απλώς αναφερόμεθα σε αυτόν. Δεν χρειάζεται λοιπόν να τα επαναλάβουμε. Νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά τεχνικής ε, της νομοθεσίας και έτσι εξασφαλίζουμε και την ε, συνέπεια με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Και κάτι άλλο που επίσης το ανέφερε η κυρία Χάουταλα. Είναι θετικό το EFSD να μπει στο εντίκι γιατί όλες οι αρχές της αποτελεσματικότητας, της βοήθειας, ε, της ε, προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, όλα αυτά θα εφαρμόζονται σε ολόκληρο το μέσο. Είτε είναι επιδοτήσει, είτε είναι δάνεια, είτε είναι εγγυήσει, ό,τι μορφή και να έχουν, όλες οι αρχές όλα τα κριτήρια αποτελεσματικότητα, ε, ανάπτυξης των ανθρώπων, ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλα αυτά θα ισχύουν για όλε τι περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν νοικοκυρεύουμε κάπως την ε, λειτουργία μας. Τέλος. Η κυρία Μάλετιτς αναφέρθηκε στην ισορροπία που πρέπει να υπάρχει όσον αφορά τον ανοιχτό χαρακτήρα της πλατφόρμας σε σχέση με την ε, συνέχιση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Εμείς θεωρούμε ότι η ΕΤΕ είναι λογικό συνομιλητή της Τράπεζας Επενδύσεων. Πρέπει να συνεργαστεί πολύ περισσότερο λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην καθημερινή μα εργασία, στην εργασία επί τόπου. Πρέπει να ξέρει από πολύ πιο κοντά ποιε είναι οι μακροοικονομικέ ανάγκε των χωρών στι οποίε εργαζόμεθα. Θεωρούμε λοιπόν ότι το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης εργάζεται για τον προγραμματισμό θα είναι προστιθέμενη αξία και την εργασία της ΕΤΕ. Και βεβαίως δεν υπάρχει καμία βούληση να θέσουμε εν κινδύνο την εργασία της ΕΤΕ. Όχι. Θέλουμε απλώς να αλλάξουμε κάπως τη μεθοδολογία της εργασίας της, ούτω ώστε να προσαρμοστεί λίγο περισσότερο στις ε, προτεραιότητες βιώσιμης ανάπτυξης των χωρών ε, με τις οποίες συνεργαζόμεθα. Με συγχωρείτε που μακρηγόρησα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε τόσο πολύ χρόνο ομιλίας. Ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά. Τώρα, να δώσω το λόγο στο συνάδελφό σας που είναι επικεφαλής για ε, την διεθνή συνεργασία και την πολιτική ανάπτυξη να προσθέσει κάποια σχόλια στην υπηρεσία εξωτερική δράση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω αγγλικά. Και εγώ συμφωνώ με τα σχόλια που καλωσορίζουν την γραμμοδότηση κυρίως στο σχόλιο ότι υπάρχει γενική υποστήριξη της ε, όλης αρχιτεκτονικής, ε, του Μηχανισμού Γειτονία Ανάπτυξης και Διεθνούς ε, Συνεργασίας, καθώς ενοποιεί υφιστάμενα μέσα και επιτρέπει να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε καλύτερα και σε προβλεπτές περιστάσεις. Καλωσορίζω και την έμφαση που δίνεται με τη μορφή πρότασης περισσότερων πόρων, της έμφασης που δίνεται λοιπόν στις προτεραιότητες που με σαφήνεια έχουν εντοπιστεί στην πρόταση, δηλαδή υποστήριξη στην υποσαχάρια Αφρική και στη γειτονία. Και φυσικά αυτό θα εξαρτηθεί από την ε, όλη ισορροπία που θα βρεθεί σε ό,τι αφορά τους πόρου για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όμως, από την εξωτερική σκοπιά, τουλάχιστον μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι για την πρόταση αυτή. Επίσης, υποστηρίζω ότι υπόθηκε από τον συνάδελφο από την Κομισιόν σε ό,τι αφορά την ε, πρόταση για ανώτατο όριο σε ό,τι αφορά το ποσοστό για την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Από ό,τι καταλαβαίνω, εδώ ε, κρατάμε τις υπόλοιπου πόρου του Ντίκη για την αναπτυξιακή δράση, αλλά δεν μπορούμε να προκαθορίσουμε ποια θα είναι η ορθή ισορροπία μεταξύ του 9% και του 50% αυτό θα το γνωρίζουμε μετά από τον προγραμματισμό, όταν θα γνωρίζουμε πού και τι θα επενδυθεί, τι θα πρέπει να υποστηριχθεί από την εγγύηση παραδείγματο ε, χάρη για ε, κρατικό δανεισμό και έχουμε εκεί χαμηλότερο ποσοστό το 9% ή άλλες συναλλαγές πιο επικίνδυνες όπου θα έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό εφοδιασμού. Έτσι λοιπόν η αλλε συναλλαγε πιο επικινδυνες οπου θα ισορροπία μεταξύ του 9% και του 50% θα είναι γνωστή μόνο όταν θα έχουμε μία ανάλυση που θα μας δίνει τις προτεραιότητες και τις ορθές στρατηγικές ε, για τις διάφορες χώρες και περιφέρειες. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η ανησυχία που εκφράζεται είναι ορθή, αλλά ίσως ο τρόπος που έχουμε προτείνει να έχουμε ένα καθολικό νοτοτόριο για την εγγύηση, ίσως ε, θα ε, πρέπει να το δούμε αυτό ανάλογα με το πώς θα λειτουργεί ο μηχανισμός. Και θέλω να επαναλάβω ότι το EFSD είναι ένα νέο τμήμα, καινοτόμο τμήμα της πρότασης DITSI, γιατί μας δίνει διάφορους τρόπους εγγύησης μακροοικονομική βοήθεια και επενδύσεων σε, ε, διάφορες, ε, σε ένα μείγμα πολιτικών και επίσης δίνει και μία συνέπεια στην ενεργοποίηση των πόρων. Ίσως να σχολιάσω και το θέμα της διακυβέρνησης του μηχανισμού. Ξέρουμε και από αυτή τη γνωμοδότηση, αλλά και από άλλες γνωμοδοτήσεις, σε άλλες επιτροπές, ότι υπάρχει έκκληση ισχυρή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει έναν ισχυρότερο ρόλο σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής των πόρων για την εξωτερική δράση. Βεβαίως, ε, δεν μπορούμε παρά να καλωσορίσουμε μια τέλεια λειτουργία ε, του δημοκρατικού ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όμως ταυτόχρονα θέλω να βιστήσω την προσοχή σας ε, στην ισορροπία μεταξύ των νομικά δεσμευτικών διατάξεων, παραδείγματο χάρη του πολλαπλασιασμού των καδεξιδότησης πράξεων και ίσως άλλων ε, πολιτικά, ίσως όχι νομικά, αλλά πολιτικά δεσμευτικά μηχανισμών, δηλαδή την ελεπίδρωση μεταξύ Κομισιών, Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι έχουμε πολλά παραδείγματα σε διάφορε επιτροπέ όπου ε, στην, ε, ο καθημερινός τρόπος ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων εγγυάται και την ικανότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εκφράζει συγκεκριμένη άποψη για το πώς ε, προωθούνται οι πολιτικές προτεραιότητες. Και ένα τελευταίο σχόλιο σε σχέση με το όσα είπε η κυρία Χαουτάλα. Βεβαίως και υποστηρίζουμε την αρχή το να έχουμε μια αναφορά στις ε, αρχές του ΟΣΑ και του ΙΕ για τα ανθρωπινά δικαιώματα και τις επιχειρήσεις. Νομίζω όμως ότι ο συνάδελφος το εξήγησε αυτό. Αυτή η γενική αρχή, αυτές οι γενικές αρχές εφαρμόζονται σε όλες τις συνιστώσεις ε, του Μηχανισμού γειτονία Ανάπτυξης και Διεθνούς συνεργασία. Έκανε επίση ένα σχόλιο για την οικοδόμηση ικανοτήτων για την ασφάλεια και την ανάπτυξη, κάτι που θα πρέπει να ειδωθεί ξεχωριστά. Η πρότασή μας είναι να διατηρήσουμε στον DC και μέσω του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις δράσεις που μπορούν να υποστηριχθούν μέσω του προπολογισμού. Παραδείγματο χάρη αυτό που υποστηρίχθηκε μέσω της ε, οικοδόμησης ικανοτήτων για την ασφαλεία και την ανάπτυξη. Ε, και αυτό συνεισφέρει στην ειρήνη και τη σταθερότητα. Δηλαδή αναγνωρίζεται ο συνδεσμός μεταξύ ανάπτυξης και ασφάλειας και βρίσκουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε ορθά τους σπόρους στον τομέα αυτό. Και για οτιδήποτε είναι πέραν αυτού του επίπεδου και αφορά θέματα άμυνας, έχουμε προτείνει τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού για την ειρήνη εκτός προϋπολογισμού. Τελείωσα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μάλιστα καθάρισαν όλα, μας διαφωτίσατε. Συμπρασματικά, κυρία Συγκήτρια, ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο για τα σχόλιά τους. Σε γενικές γραμμές συμφωνούμε μεταξύ των ομάδων. Μπορεί να υπάρχει κάποια μικρή απόχρωση σε σχέση με το τι είπε η κυρία Χαουτάλα εγώ δεν έχω παρουσιάσει τροπολογίες προς αυτήν την κατεύθυνση, όχι επειδή δεν είχα διάθεση, αλλά γιατί προσπάθησα να περιοριστώ στο διονυμοσιονομικό σκέλος ε, αυστηρά. Όμως ε, με την παράτιμη μετανάστευση και με την πολιτική του φίλου δεν μπόρεσα να αντισταθώ και εκεί παρουσίασα κάποιες τροπολογίες. Άλλος αυτός ο μηχανισμός ε, μπαίνει υπό την πολιτική συνεργασίας όμως πολλές φορές καλύτερα είναι ε, να έχουμε επικάλυψη αν ε, και δεν είναι πολύ υγιές να το κάνουμε αυτό από νομοθετική σκοπιά, αλλά πολιτικά καλύτερα να παραλάβουμε δύο φορές την ίδια ιδέα παρά να την ξεχνάμε σε ό,τι αφορά τώρα τον αφοδιασμό της εγγύησης, εγώ καταλαβαίνω, καθώς έχουμε διάφορους ε, πρώην μηχανισμούς, κατανοώ το να το αφήσουμε ανοιχτό και να πρέπει να αφοδιάσουμε από το 9% μέχρι το 50% ανάλογα με το είδος ε, της ε, πράξης. Και καθώς δεν ξέρουμε τι θα χρειαστεί, πρέπει να το αφήσουμε ανοιχτό. Όμως, νομίζω ότι να το αφήσουμε τόσο ανοιχτό μπορεί να έχει κάποιους κινδύνους. Γι' αυτό θεωρούσα αρκετά λογικό να βάλουμε αυτό το σημείο ελέγχου, δηλαδή χρειαζόμαστε να ενεργοποιήσουμε πάνω από 10 δισεκατομμύρια για την εγγύηση, να το δούμε, να το συζητήσουμε και να το υιοθετήσουμε. Και γι' αυτό εγώ θεώρησα ότι είναι σημαντικό να έχουμε αυτό το σημείο ελέγχου, δηλαδή όχι να έχουμε έλλειψη ευελιξίας, αλλά να κάνουμε ακριβώς αυτό που πρέπει και να μην πηγαίνουμε σε ε, υπερβολικούς κινδύνους. Τώρα για τη συμμετοχή. Ήταν κάτι επίμαχο και όταν είχαμε τις συζητήσεις για το προηγούμενο Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι προτάσεις οδεύουν προς το να διευρυνθεί συμμετοχή άλλων εντοτήτων στη χρήση της εγγύησης αυτής. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όχι μόνο είναι σε πλήρη θέση και ικανή να χρησιμοποιήσει αυτή την εγγύηση, αλλά είναι αυτό που καλύτερα έχει κάνει και θα κάνει ε, με την εντολή εξωτερικού δενισμού Και ωστόσο η ΕΤΕ θα πρέπει ε, να υλοποιήσει αυτή την ε, εντολή και δεν χρειάζεται εμείς να βάλουμε κάποια σχετική διάταξη γιατί είναι ειδική η ΕΤΕ σε τέτοιο είδου προγραμματισμό. Όμω είχαμε συνεδριάσει για αυτό το θέμα και ξέρω ότι και η Κομπισιόν γνωρίζει ότι υπάρχει ένας φόβος στην ε, μετάβαση από το External Lending Mandate σε αυτό το νέο μηχανισμό. Και λόγω αυτής της μετάβασης και λόγω των διάφορων τεχνικών προβλημάτων που προέρχονται από την υποχρέωση υπογραφής νέων συμβάσεων μπορεί να υπάρχει μια περίοδος όπου υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να χαθεί χρηματοδότηση θα πρέπει να εργαστούμε σε αυτό. Εγώ δεν έχω την ε, τεχνική ικανότητα να σκεφτώ πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και ίσως ε, στην Κομπισιόν ή στο Συμβούλιο να υπάρχουν εμπειρογνώμες που να μπορούν να το κάνουν αυτό. Βέβαια, ξέρω ότι υπάρχει αυτός ο φόβος. Και δεν έχω κάποια σχετική πρόταση. Όμως ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε να γίνει αυτή η μετάβαση για να μην σταματήσουν να γίνονται τέτοιες συναλλαγές ε, που σχετίζονται με το external lending mandate. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποια περαιτέρω διάταξη και είναι υγιές οι οντότητες που μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό, να συνεργαστούν ε, και ίσως και να συναγωνιστούν, γιατί έτσι θα έχουμε τους ειδικού από κάθε μηχανισμό, από κάθε περιοχή και από κάθε πρόγραμμα που θα υλοποιούν ε, την ε, δραστηριότητα αυτή. Αυτά από μένα και περιμένω τις τροπολογίες σας. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα πρέπει λοιπόν ταυτόχρονα να είμαστε τολμηροί αλλά και σόφρονες. Όταν δεν έχουμε χρήματα είναι πολύ ωραία η μηχανική ε, γιατί ουσιαστικά έχει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Στην αρχή όλα πάνε καλά, τα πρώτα χρόνια, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά προσοχή. Είμαστε εδώ σε ένα έδαφος που δεν μπορούσαν να εξαφανιστούν πολύ γρήγορα επιστώσεις. Έτσι λοιπόν, να μην υποτιμάμε τον κίνδυνο που αναλαμβάνουμε και να προσπαθήσουμε τα κονδύλια για την εγγύηση να τα διατηρούμε σε ένα προληπτικό επίπεδο. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να σας διευκρινίσω, αφού ευχαριστήσω εκ νέου την συγγήτρια, ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι στις 26 Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, την επόμενη Δευτέρα. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 10 Δεκεμβρίου. Η Κοινή Επιτροπή ΑΦΕΤ και ΝΤΕΒΕ θα ψηφίσει στις 4 Φεβρουαρίου και ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα έχουμε στις 11 Φεβρουαρίου. Τώρα έχουμε την έκθεση του κυρίου Κέλμελ για την ε, απλούστευση του συστήματος χορήγησης θεωρήσεων. Ο κύριος ε, Κέλμελ έχει καταρτήσει τη γνωμοδότηση και έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, εδώ μιλάμε για το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το όλο σύστημα έχει ως εξής. Η Κομισιόν υποβάλλει πρόταση τροποποίησης διαφόρων άλλων πράξεων και ε, ε, επί της αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή ΛΥΜΠ, εμείς γνωμοδοτούμε. Από άποψη περιεχομένου, η πρόταση της Κομισιόν είναι εξαιρετική. Γιατί πράγματι γνωρίζουμε ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμούν πολύ την ελευθερία κυκλοφορίας και ε, όχι μόνο ε, οι πολίτες μας και οι επιχειρήσεις χρειάζονται αυτή την ελευθερία. Οτιδήποτε άλλο θα, τη ζημίωνε, θα ζημίωνε τις επιχειρήσεις σημαντικά. Για να μπορεί όμως να εξασφαλιστεί αυτή η ελευθερία κυκλοφορίας εντός του Σέγγεν θα πρέπει να προστατεύονται με τέτοιον τρόπο τα εξωτερικά σύνορα ώστε αυτός ο χώρος ελευθερίας να μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει. Και σε αυτό βεβαίως συγκαταλήγεται και ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις. Με τις προτινόμενες αλλαγές, οι έλεγχοι στα σημεία διέλευσης των συνόρων απλουστεύονται, αλλά και ενισχύονται ταυτόχρονα. Σκοπός είναι να υπάρξει καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόστροι των χωρών, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους θεώρηση ή άδεια διαμονής ε, μακρόχρονης διάρκειας. Όλα αυτά είναι απαραίτητα πλέον σήμερα και για να εξασφαλιστεί κάτι τέτοιο χρειάζεται βεβαίως και πληροφοριακό σύστημα. Χωρίς πληροφορικά συστήματα δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα. Γι' αυτό αναγκαίο είναι να γίνουν επενδύσεις. Συνολικά μιλάμε για 182 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά τα χρήματα και μιλάμε συγκεκριμένα για 105 εκατομμύρια ευρώ για τον Ιουλίζα, 45 εκατομμύρια ευρώ για τα κράτη-μέλη που θα μεταφέρουν τα χρήματα αυτά στα εθνικά τους προγράμματα, 2 εκατομμύρια ευρώ για τον Frontex και 30 εκατομμύρια ευρώ για την Ευρωπόλη. Όπως είπα, το ποσό είναι μεγάλο. Εμείς δεν έχουμε ε, πληροφορίες για το ότι θα μπορούσε να είχε διαμορφωθεί το κόστος και σε χαμηλότερα επίπεδα. Γι' αυτό και απλά ε, τους πιστεύουμε. Δεν έχω όμως και κανένα λόγο να πιστεύω το αντίθετο. Είναι δικαιολογημένα τα κόστη αυτά, διότι σε αυτού σε αυτούς τους τομείς χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις και το αξίζει η ασφάλεια των πολιτών μας. Από αυτή την άποψη δεν έχουμε και ε, επί της ουσίας ε, παρατηρήσεις να κάνουμε για την έκθεση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Ωστόσο θα υποβάλουμε κάποιες λίγες ε, τροπολογίες που ενισχύουν την κοστοποδοτικότητα, ε, και ενισχύουν τους ελέγχους των προγραμμάτων όσον αφορά την επίτευξη των στόχων από πλευράς τους ε, και την, ε, τον εξορθολογισμό του, τον, του κόστους. Διότι όταν μιλάμε για τόσα μεγάλα ποσά, προφανώς χρειάζεται και η αντίστοιχη εποπτεία και παρακολούθηση ανα πάσα στιγμή. Γι' αυτό και σας παρακαλώ εμείς ως Επιτροπή Προλογισμών να εγκρίνουμε τη γνωμοδότησή μου. Κατά τα άλλα ε, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με το συνολικό περιεχόμενο της έκθεσης. Ευχαριστώ κύριε Κόλμελ. Η κυρία Κλόντια Ταμπαρντέλ, ε, Σκιώδης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο, τον κύριο Κολμέλ, για την έκθεση. Βλέπω ότι θέλει να διατηρήσει τις δημοσιονομικές πτυχές. Εγώ υποστηρίζω αυτή την ιδέα. Επίσης, υποστηρίζω τον ε, εισηγητή ότι αντικατρίζονται αυτέ οι πτυχέ ε, καθώ και ενδυνάμωση κάποιων προβλέψεων ε, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση και την υποβολή εκθέσεων και να διασφαλίσει ότι αρμόδιε αρχέ μπορούν να παρακολουθούν εκ του σύνοικη τη λειτουργία και την πηγήτηση του συστήματο ΒΙΣ. Κατά την άποψή μου όμω θεωρώ ότι για να διασφαλίσουμε την ε, ε, πλήρη λειτουργία του συστήματος προστασίας και ελέγχου των συνόρων. Ε, οι ταξιδιώτες που έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς ελέγχου στα σύνορα θα πρέπει η Βουλγαρία και η Ρουμανία να γίνουν πλήρη μέλη του χώρου Σέγγεν, έχοντας κατά νου ότι και η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο έχουν τοποθετηθεί θετικά σε σχέση με το οι δύο χώρε Βουλγαρία και Ρουμανία πληρούν όλε τι απαραίτητε προϋποθέσεις για να αποτελούν πλήρη μέλη του χώρου Σένκεν. Θα ήθελα να θέσω αυτή την πτυχή και ελπίζω ότι θα μπορέσω να έχω και την υποστήριξη των συναδέλφων από την Ευρωπαϊκή Προϋπολογισμών, αν και αυτό δεν είναι ένα συγκεκριμένο θέμα που πάπτεται των αρμοδιοτήτων σα. Όμω νομίζω ότι για την καλύτερη λειτουργία αυτού του συστήματο, ε, χρειαζόμαστε να ενταχθούν όλα τα κράτη-μέλη στο χώρο Σέγγεν. Επίσης, καθώς συζητάμε για ολοκληρωμένα συστήματα ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, ακριβώς για να ενισχύσουμε τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα, μου φαίνεται αφύσικο δύο από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται στα ανατολικά ε, εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην είναι πλήρη μέλη του χώρου Σέγγεν, καθώς μάλιστα πληρούν όλα τα τεχνικά κριτήρια για να είναι μέλη αυτού και συμμετέχουν μάλιστα και σε όλα τα συστήματα πληροφορικής υποβολής εκθέσεων σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των συνόρων. Θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Εγώ θα υποστηρίξω την προσέγγιση του κυρίου Κέλμα, αλλά θα υποστηρίξω και αυτή την κατεύθυνση που σας ανέφερα και έχω την πεποίθηση ότι θα φτάσουμε σε συμβιβασμούς που να συμπεριλάβουν και την πτυχή της οποίας, την οποία σας ανέφερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, δεν βλέπω να θέλει λόγο. Α, είσαστε τόσο πολύ με στην αίθουσα. Φαίνεται ότι τα επιχειρήματα του εισηγητή σας έπεισαν. Κύριε Κόλμελ, για να ολοκληρώσετε αυτή την ανταλλαγή απόψε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με δύο λόγια θέλω να ευχαριστήσω την συνάδελφο για την παρέμβασή της. Συμφωνώ μαζί της. Αν θέλουμε να έχουμε ένα χώρο Σέγγεν, αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα το αν η συγκεκριμένη έκθεση είναι ο κατάλληλος χώρος όπου μπορούμε να επαναλάβουμε το αίτημά μας αυτό επιτακτικά, δεν το ξέρω. Ίσως ε, εξαρτάται και από τη διατύπωση. Γιατί όχι να υπάρχει μια παραπομπή σε αυτό το θέμα ε, πάντως ε, σε κάθε περίπτωση πρέπει να πάρουμε τα μέτρα ε, τα απαραίτητα προκειμένου να ευοδοθεί αυτό το αίτημα και να πράγματι να ενταχθούν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χώρο Σέγγεν. Ο χώρο Σέγγεν είναι σαν την Ευρωζώνη. Όλες οι χώρες μπορούν να ενταχθούν. Αυτά γι' αυτό. Την τροπολογία σας παρακαλώ, κυρία μου μέχρι τις 12 ώρα τη 27 Η Νοεμβρίου. Ε, όχι μόνο, εσείς βεβαίω και όσοι άλλοι ενδεχομένω θέλουν. Η Επιτροπή Προπολογισμών θα ψηφίσει στις 23 Ιανουαρίου και η ΛΥΜΠΕ επίση τον Ιανουάριο. Δηλαδή στις 8 μέρες που απομένουν στο μήνα. Και τώρα ο Ζωζέ Μανουέλ Φερνάνδες, μέγας ειδικό για θέματα αλίας, για την ε, συμφωνία αλίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Στην έκθεση αυτή, στην έκθεση γνωμοδότησης, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν τροπολογίες και απλώς ε, μπορούμε να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας, ε, ναι ή όχι. Και ε, μερικές ε, φορές ε, η ερώτηση αν είναι κάτι πολύπλοκο και η απάντηση είναι ή όχι. Δεν θα υπάρχει λοιπόν δυνατότητα κατάθεσης τροπολογιών. Η αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Αλίας η οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σχέση με όλες ε, τις ε, πολιτικές ε, πτυχές και σε σχέση με όλο το φάκελο από δημοσιονομική σκοπιά. Εμείς, εγώ είμαι υπέρ για τη συμφωνία αυτή ετήσια η χρηματική αντιπεροχή έχει οριστεί στα 37 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε μία ετήσια αύξηση μέχρι να φτάσει το τελευταίο έτος στα 42,4 εκατομμύρια ευρώ. Στο τέταρτο έτος ε, θα φτάσουμε εκεί γιατί η συμφωνία προβλέπει τη διάρκεια των τεσσάρων ετών. Όπως ε, σας είπα, ε, δεν είναι αποκλειστική δική μα αρμοδιότητα. Αρμόδια είναι η Επιτροπή Αλία. Όμω, ε, εγώ είμαι θετικό απέναντι στη συμφωνία γιατί λαμβάνει υπόψη όλο τον πληθυσμό και όλη την προβληματική που υπάρχει στην ε, περιοχή. Και έχουμε εδώ σκοπό να βοηθήσουμε όλον τον πληθυσμό έχουν απαντηθεί και οι ανησυχίε μας για μια ελία που πρέπει να είναι φιλική προς το περιβάλλον. Η δική μου έκθεση λοιπόν έχει μια πολύ σύντομη αιτιολόγηση. Δεν μπαίνουμε στην ανάλυση επί της ουσίας. Εδώ προτείνω να έχουμε θετική απάντηση από τη δική μας πλευρά και στη συνέχεια να αποφασίσει η Αρμόδια Επιτροπή, που είναι η Επιτροπή Ελίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκαρδιά Σαβάλ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Έχει μείνει ο εισηγητής και εγώ και ο πρόεδρος. Νομίζω ότι αν συμφωνεί και ο πρόεδρος ε, θα υπήρχε απόλυτη ομοφωνία με τον εισηγητή και αν συμφωνούμε και οι τρεις μας. Στηρίζω λοιπόν τη σύμφωνη γνώμη προς την συμφωνία με το Μαρόκο. Οι συνάδελφοί μας έχασαν ε, μια θαυμάσια συζήτηση. Α, τιμωρούνται. Νομίζω ότι υπάρχει γενικά συνένεση. Και δεν νομίζω ότι οφείλεται στην κούραση άριστα. Μετά αυτή την πλούσια ανταλλαγή απόψεων όσοι έχουν αντίρρηση σε αυτή τη συνένεση μπορούν να υποβάλουν τροπολογίες. Και αν προτίθεται να το κάνουν θα πρέπει να το κάνουν ε, μέχρι τις 12 η ώρα της 23ης τρέχοντος. Θα ψηφίσουμε στις 10 Δεκεμβρίου θα δώσουμε κατά πάσα πιθανότητα τη σύμφωνη γνώμη, οπότε δεν θα υπάρχουν τροπολογίε. Δεν θα μπορούν να γίνουν δεκτέ τροπολογίε. Η Επιτροπή Αλία θα ψηφίσει 23 Ιανουάριου και η Ολομέλεια το Φεβρουάριο. Διάφορα. Έχει κανείς διάφορα. Όχι. Οπότε η επόμενη, οι επόμενες συνεδριάσεις μας θα γίνουν στις 26 Νοεμβρίου μαζί με την Μπάτζ και την ΕΚΟΝ αλλά πρέπει ακόμη να επιβεβαιωθεί στις 27 Νοεμβρίου α όχι άλλο, στις 27 Νοεμβρίου 10 και 10.45 Μπάτζ ΕΚΟΝ για θέματα των τροπολογιών για την λειτουργία σταθεροποίησης. Είναι συνέχιση της έκθεσης Burger Μπέρες. 27 Νοεμβρίου επίσης. 27 Νοεμβρίου. Μια κοινή συνεδρίαση λοιπόν Badge Cont και ημών για το κράτος δικαίου. 3 Δεκεμβρίου. Μποτζεκόν, Παρουσίαση της δεύτερης εκδοχής ενδεχομένως του προπολογισμού 2019 με τουλάχιστον 150 εκατομμύρια για την έρευνα με εφαρμογή του 15-3 10 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο και στις 13 Σεπτεμβρίου, ε, Δεκεμβρίου Μποτζεκόντ. Και αυτό θα ικανοποιήσει ιδιαίτερα την Γαλλία, γιατί δεν ήθελε η ψηφοφορία να γίνεται στι Βρυξέλλε για τον προπολογισμό. Αυτή τη φορά, βεβαίω, αν υπάρξει συμφωνία, θα ψηφιστεί στο Στρασβούργο ο προπολογισμό. Εάν δεχθούν όμω το 15-3. Αλλιώ θα ψηφιστεί τον Ιανουάριο, στο Στρασβούργο όμω. Να προειδοποιήσετε λοιπόν την Ρουμανική Προεδρία. Άριστα. Καλά περάσαμε. Ευχαριστώ τους συμμετέχοντες, ευχαριστώ την γραμματεία μας, ευχαριστώ τους διερμηνείς, ευχαριστώ τους ε, πολιτικούς συμβούλους, σας ευχαριστώ όλους κύριε και κύριοι και με χαρά θα τα ξαναπούμε. Καλό σας βράδυ. Λήξη τη συνεδριάσεως.